Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα παρακαλώ να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Οι Δευτέρες είναι πάντα δύσκολες μέρες. Πολλοί συνάδελφοι έχουν και άλλες ενηλυμένες υποχρεώσεις στις εκλογικές τους περιφέρειες και δεν προλαβαίνουν όλοι να έρθουν εγκαίρως για τη συνεδρίασή μας Δευτέρα απόγευμα. Αλλά αυτό είναι τμήμα του κοινοβουλευτικού έργου, να αφιερώνει ένα τμήμα του χρόνου ο Ευρωβουλευτής και στους ψηφοφόρους του. Η σημερινή μερίσια διάταξη σας έχει μοιραστεί. Δεν βλέπω παρατηρήσεις, οπότε μπορούμε να την εγκρίνουμε ως έχει. Αναμεταδίδεται και από το διαδίκτυο η συνεδρίασή μας και έχουμε σε 20 γλώσσες διερμηνία με εξαίρεση τα μαλτέζικα, σλοβακικά και εγωεδελικά. Ως ήθιστε θα ήθελα να εγκρίνουμε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 21ης και 25ης και 26ης Απριλίου. Και περνάμε στο σημείο 4, την παρουσίαση της μελέτης με θέμα η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα μέσα διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη κατά την περίοδο 2014-2020 εθνικά και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχουμε ε, τη μελέτη που έγινε με το συντονισμό του Ερευνητικού Κέντρου για τη Διαχείριση της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος και των σχετικών κινδύνων και με συνεργασία με διάφορους φορείς από τη Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, δηλαδή το Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, στις Αλπ, στην περιοχή Αλπ, των Άλπαιων, ε, το Πανεπιστήμιο της Νάπολης και το Ινστιτούτο Οικονομίας, Γεωγραφίας και Δημοκρατίας της Μαδρίτης. Όλοι αυτοί οι φορείς συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης, της μελέτης. Η μελέτη έχει στόχο την ε, αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν εφαρμόσει τα κράτη-μέλη για να διαχειριστούν τον κίνδυνο στον γεωργικό τομέα, τους κινδύνους στον γεωργικό τομέα. Αυτό είναι το αντικείμενο της μελέτης η μελέτη αναλύει τι ομοιότητε και τι διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη χρήση μηχανισμών και εργαλείων για τη διαχείριση των κινδύνων. Και είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της χρήσης αυτών των μηχανισμών. Και επίσης από τη μελέτη θα προκύψουν και κάποιες συστάσεις για την μελλοντική πορεία της κοινής γεωργικής πολιτικής και την αξιοποίηση διαφόρων μέσων για τη διαχείριση των κινδύνων στην κοινή ιωρική πολιτική. Η μελέτη αφορά ένα σημαντικό θέμα και ευαίσθητο πως είναι η αβεβαιότητα ως προ το γεωργικό εισόδημα, αλλά και η αστάθεια στις γεωργικές αγορές. Οι ε, καλεσμένοι μας είναι εμπειρογνώμονες. Η κυρία Ισαμπέλ Μπαρντάη από το Ερευνητικό Κέντρο για τη Διαχείριση των Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων από την Ισπανία. Ο κύριος Χωσέ Μαρία Σούμψη από το ίδιο Ερευνητικό Κέντρο, το ΣΕΙΚΡΑΜ της Ισπανίας. Και ο κύριος Τόμας Γκαρσία Ασκαράτε από το Ινστιτούτο Οικονομίας, Γεωγραφίας και Δημογραφίας της Ισπανίας. Την παρουσίαση θα μας την κάνει η κυρία Μπαρντάγιχη και κατόπιν ε, θα γίνει συζήτηση με υποβολή απορριών και ερωτήσεων. Σίγουρα θα υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις, στις οποίες θα απαντήσουν και οι τρεις εμπειρογνώμονες ε, που έχουμε προσκαλέσει. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την κυρία Μπαρταχή να μας κάνει την παρουσίαση. και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω αυτή τη μελέτη που έγινε με ανάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα αναφερθώ πρώτα απ' όλα στους στόχους αυτής της μελέτης, σε συντομία στο πλαίσιο στήριξη, στον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ενίσχυσης, των μέτρων στήριξης θα αναφερθώ στην εφαρμογή των μέτρων στήριξης από τα κράτη-μέλη. Θα σας παρουσιάσω κάποιες κέρυες ιδέες που θα αποτελέσουν και τη βάση των συστάσεων που θα σας κάνουμε για το τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο σύστημα στήριξης των μέσων διαχείρισης κινδύνων και θα ολοκληρώσω με κάποια συμπεράσματα και συστάσεις. Καταρχήν, ποιοι ήταν, ήταν οι στόχοι της έκθεσης. Η της μελέτης. Η μελέτη είχε ως στόχο την ανάλυση της χρήσης των διαφόρων μέσων στήριξης ε, για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στα κράτη-μέλη και το πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα μέσα στήριξης. Και ανάλογα με τα αποτελέσματα, δεύτερο στόχος της μελέτης μας ήταν ε, να προτείνουμε πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο στήριξης αυτών των μέσων διαχείρισης κινδύνων το πλαίσιο στήριξη ε, των μέσων διαχείριση κινδύνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται από τους κανόνε ε, της Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Αυτά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της Συμφωνία τη Γεωργίας, ε, που προβλέπει τι διατάξει θα πρέπει να ισχύουν για τα μέσα διαχείριση κινδύνων, ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν ω πράσινο κουτί και να θεωρούνται αποδεκτά στα πλαίσια αυτού του πλαισίου. Αφορούν δύο πτυχές αυτές ε, οι διατάξεις. Καταρχήν, τις ασφαλίσεις ε, ε, εισοδήματος και ασφαλών δικτύων εισοδήματος και εξασφάλιση των συγκομιδών. Για να είναι μια ενίσχυση ενίσχυση του πράσινου κουτιού θα πρέπει η απόλυση ζημίας να είναι πάνω από 30% του μέσου εισοδήματος των τριών τελευταίων χρόνων, η ε, αντιστάθμιση λιγότερη από 70% της απώλειας του εισοδήματος και αυτή η αποζημίωση να σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με το εισόδημα, ούτε με τις ε, τιμές, ούτε με την παραγωγή, ούτε με το κόστος της παραγωγής. Σε ό,τι αφορά τις ε, ασφάλειες εσοδείας, καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει επίσημη αναγνώριση της θεομηνίας για να επιτρέπεται αποζημίωση. Θα πρέπει οι ζημίες να είναι μεγαλύτερες από το 30% της μέσης παραγωγής των τριών τελευταίων χρόνων. Οι πληρωμέ ή οι αποζημιώσει να σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τι ζημίε που έχει προκαλέσει η σχετική θεομηνία ή η φυσική καταστροφή και θα πρέπει οι επιζημιώσει αυτέ να αντικαθιστούν, να είναι μεγαλύτερε από την αντικατάσταση του κόστου ε, τη θεομηνία και να μην σχετίζονται με την παραγωγή. Αυτοί είναι οι κανόνε που προβλέπει η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορική είναι αρκετά περιοριστικοί αυτοί οι κανόνες ε, για το τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μία διάταξη, ένα μέσο για να εμπίπτει στο πράσινο κουτί. Τώρα, πώς δρομολογείται αυτή η στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται διάκριση μεταξύ δύο περιόδων περίοδου 2007-2013 και της ε, τωρινής περίοδου 2014-2020. Στην πρώτη περίοδο, 2007-2013, οι δυνατότητες που είχε ένα κρατός μέλος για να στηρίξει τα μέσα διαχείρισης κινδύνων ή κρίσης ήταν καταρχήν η κρίση ηταν καταρχην γεωρική πολιτική με το άρθρο 68 του κανονισμού της ενιαίας ενίσχυσης και κάποιες ειδικές προϋποθέσεις για οποροκυπευτικά και ίνο. Έχουμε όμως και τη δυνατότητα των κρατικών ενισχύσεων. Κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπουν ε, τους όρους από τους οποίους επιτρέπονται οι κρατικές ενισχύσεις αφορούν δύο πτυχές. Καταρχήν, οι εκ των προτέρων ενισχύσεις, που είναι επιδοτήσεις και ασφάλειες ε, της τα ή βέα κεφάλαια, ή εκ των υστέρων ε, ενισχύσεις, που προβλέπουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ε, χορηγούνται ad hoc ενισχύσεις. Αυτό το πλαίσιο στην παρούσα περίοδο έχει αλλάξει. Κυρίω ό,τι αφορά τα μέσα στήριξη διαχείριση κινδύνων ε, εντό τη κοινή γεωργική πολιτική. Διατηρείται η ειδική στήριξη των απορροκυπευτικών και του ίνου, αλλά η στήριξη στα μέσα ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, ασφάλεια ε, εσοδίας και αμοιβαίων κεφαλών πέρασε από πέρασαν από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Αυτή είναι η πιο σημαντική αλλαγή. Και ε, ισχύουν και πάλι προϋποθέσεις για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, εξάντα και εξπόστ. Αυτό το πλαίσιο είναι πολύ ελαστικό, θα το δούμε και στη συνέχεια, και επιτρέπει την προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρατών μελών και στην αναμοιομορφία που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών και οδήγησε στην ανάπτυξη πολύ διαφορετικών μοντέλων μεταξύ των κρατών μελών η στήριξη στην ΚΑΠ πέρασε από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα με συνέπειες που αφορούσαν τα ειδικά χαρακτηριστικά των δύο πυλώνων και το βασικό είναι ότι η βασική ενίσχυση της ΚΑΠ είτε το άρθρο 68 στην προηγούμενη περίοδο ή ο πυλώνας 2 είναι δυνατή αυτή η προσφυγή μόνο εφόσον πρόκειται για ενίσχυση στα πλαίσια του πράσινου κουτιού, δηλαδή για πολύ σημαντικές ζημιές πάνω του 30% ε, της παραγωγής ή του εισοδήματος. Οπότε είναι δυνατότητα σε τέτοιε περιπτώσει να χρησιμοποιηθούν κρατικέ ενισχύσει για μέσα διαχείριση κινδύνου που καλύπτουν ε, λιγότερο μεγάλε ζημίε, κάτω του 30%. Σε ό,τι αφορά την κάλυψη ε, κινδύνων αγορά, για πρώτη φορά συμπεριλήθηκε στο ισχύον μέσο ε, πλαίσιο στήριξης 2014-2020 με το μέσο σταθεροποίηση εισοδήματο. IST. Είναι το μόνο μέσο που επιτρέπεται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του κοινοτικού πλαισίου για την κάλυψη κινδύνων αγορά και επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια αμοιβαίων κεφαλαίων. Τώρα, πώς εφαρμόστηκε, να δούμε μερικά στοιχεία. Καταρχήν αυτό που επιτρέπει το πλαίσιο είναι μια μεγάλη ποικιλομορφία των μέσων που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη και πολυμορφία. Το άρθρο 68 της κοινή ιωρική πολιτικής χρησιμοποιήθηκε μέχρι στιγμής μόνο από την ε, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία και κατοχώρες και μάλιστα για μικρά ποσά που αφορούσαν τι ασφαλίσεις. Η στήριξη αμοιβαίων κεφαλαίων δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετά και ιστορικά οι ποσότητε ήταν πολύ μικρέ, δεν χρησιμοποιήθηκε δηλαδή το μέσο των αμοιβαίων κεφαλαίων ιδιαίτερα, ενώ όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν τι κρατικέ ενισχύσει ε, σε διαφορετικό βαθμό βέβαια ή τα άλλα μέτρα στήριξη. Τώρα, εδώ έχουμε την τυπολογία στην εφαρμογή των μέτρων στήριξης. Έχουμε την, την κατανομή των κρατών μελών ανάλογα με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκαν, είτε μέσω της ΚΑΠ είτε μέσω των κρατικών ενισχύσεων. Όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν είτε την ΚΑΠ είτε τις κρατικές ενισχύσεις για να στηρίξουν είτε τα εξάντε μέτρα, δηλαδή στηρίξη ασφαλίσεων και αμοιβαίων κεφαλαίων, είτε για την παροχή ad hoc ενισχύσεων. Αυτό φαίνεται καλύτερα σε αυτό το πίνακα, με στοιχεία που προβλέπει τις δημόσιες δαπάνες σε μέσα διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων για την περίοδο 2007-2013. Εδώ περιλαμβάνονται όλα τα κράτη-μέλη. Στην πρώτη στήλη έχουμε τα κονδύλια που αφιερώθηκαν στις εκ των υστέρων ε, ενισχύσεις διαχείρισης των ε, κρίσεων, μετά ad hoc ενισχύσεις και εξάντε ε, ενισχύσεις για τη διαχείριση των κινδύνων. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε. Αν περιοριστούμε στα τελικά στοιχεία του τελευταίου καταλόγου, βλέπουμε ότι τα 14 δις 482 εκατομμύρια, το μεγαλύτερο τμήμα προέρχεται από κρατικέ ενισχύσει. Και εντό των κρατικών ενισχύσεων έχουμε κυρίω ad hoc ενισχύσει για τη διαχείριση των κρίσεων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό. Απορροφήθηκε από αυτά τα μέσα. Τα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί από χρήματα τη κοινή γεωργική πολιτική είναι πολύ λιγότερα. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι όσο μεγαλύτερη ήταν οι δαπάνες ε, εκ των προτέρων μέτρα, τόσο μικρότερες ε, ε, δαπάνες χρειάστηκε αργότερα, χρειάστηκαν αργότερα για ex post μέτρα. Όσο, δηλαδή, όσο περισσότερα κονδύλια δόθηκαν για τη διαχείριση των κρίσεων, τόσο λιγότερα χρειάστηκαν για τη διαχείριση των κρίσεων αργότερα. Τώρα, πώς άλλαξε αυτό το πλαίσιο από την πρώτη περίοδο 2007-2013 στη δεύτερη 2014-2020. Εντός της κοινή γεωρικής πολιτικής είχαμε κάποιες μικρές αλλαγές, όχι εντυπωσιακέ. Καταρχήν να βλέπουμε στην ΚΑΠ τι έκαναν τα κράτη-μέλη και οι χώρες που χρησιμοποίησαν το άρθρο 68, δηλαδή Ιταλία, Γαλλία, Ουγγαρία και Ολλανδία. Οι χώρες αυτές ε, χρησιμοποίησαν τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου, του δεύτερου πυλώνα, και σε αυτές τις ε, τέσσερις χώρες προσθέθηκαν και άλλες που όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν κονδύλια της κοινή διορικής πολιτικής για μέσα στήριξης α, ε, διαχείρισης των κινδύνων. Και πάλι τα αμοιβαία κεφάλαια δεν στη, στηρίζονται ιδιαίτερα. Και το θέμα της σταθεροποίησης εισοδήματος χρησιμοποιήθηκε μόνο από την Ιταλία, Ουγγαρία και η Ισπανία και κυρίως από την Καστίγια Λεόν, αυτή την περιοχή της Ισπανίας. Και εδώ βλέπουμε τις ταπάνες που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια των προγραμμάτων ανάπτυξη υπαίθρου για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού. Και βλέπουμε πως κάποιες χώρες που ήδη ξεκίνησαν να εισάγουν την στήριξη ασφάλισης ε, στα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου και Μόνο η Καστίγια, η Λεόν από την Ισπανία, η Ιταλία και η Ουγγαρία είτε διατηρούν είτε θεσπίζουν τη δυνατότητα του μέσου σταθεροποίησης εισοδήματο. Κάτι άλλο που βλέπουμε είναι το σύνολο της ε, ενίσχυσης που έχει προγραμματιστεί για τα μέσα διαχείρισης ε, κινδύνων. Είναι 2 ε, δις 700 εκατομμύρια την περασμένη περίοδο είχαμε 800 εκατομμύρια. Η αλλαγή είναι αρκετά σημαντική. Και βέβαια σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις είναι πολύ μικρότερο το ποσό, αλλά όλο και περισσότερες χώρες στηρίζουν, αρχίζουν και στηρίζουν κάποια μέσα διαχείρισης των κινδύνων. Εδώ έχουμε, πέραν των κρατικών ενισχύσεων, κάποια μέσα διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων βλέπετε ότι οι τάσεις διατηρούνται, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, δηλαδή οι αλλαγές είναι σχετικά άτολμες και διατηρείται η διαφορετική χρήση των εφιστάμενων μέσων από τα κράτη-μέλη. Εδώ έχουμε κάποιες ε, βασικές ιδέες που μπορούν να χρησιμεύσουν για τον καλύτερο σχεδιασμό των μέσων διαχείρισης κινδύνων. Σε αυτή την πυραμίδα βλέπουμε την κατανομή των κινδύνων ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. Στη βάση της πυραμίδας έχουμε τους κινδύνους που αναλαμβάνει ο γεωργός ή μια οργάνωση παραγωγών, χωρίς να χρειάζεται μετακύληση του κινδύνου ή μεταφορά του κινδύνου. Εδώ μιλάμε για κινδύνους που κάλλιστα θα μπορούσε να τις αναλάβει μέσω ιδιωτικής διαχείρισης ο Γεωργός ή με τη διαφοροποίηση κάποιων μέτρων για τις οργανώσεις παραγωγών. Και είτε οι ίδιοι παραγωγοί είτε οι οργανώσεις τους αναλαμβάνουν αυτό το πρώτο επίπεδο, το πρώτο στρώμα κινδύνου. Στο μέτρο όμως που αυξάνεται ο κίνδυνος, περνάμε σε άλλα μέσα διαχείρισης κινδύνων. Εκεί έχουμε μια μεταφορά, μετακύληση του κινδύνου από τον Γεωργό σε κάποιο τρίτο. Και εδώ έχουμε τις ασφαλίσεις ή τα αμοιβαία κεφάλαια. Εδώ έχουμε διαφορετικά μέσα και μηχανισμούς ανάλογα με την κάλυψη των ζημιών και πόσο σοβαρές είναι αυτές οι ζημίες. Και επίσης αυτά τα μέσα θα χρηματοδοτούνται από κοινού από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και περνάμε στην κορυφή της πυραμίδας που είναι ο καταστροφικός κίνδυνος, οι μεγάλες κρίσεις ε, και ο κίνδυνος αυτός αναλαμβάνεται κυρίως από δημόσια χρηματοδότηση. Το σημαντικό στην πυραμίδα αυτή είναι να θεωρήσουμε ότι όλοι οι κίνδυνοι θα πρέπει να εξεταστούν σε διάφορα στρώματα. Υπάρχει μια διαστρωμάτωση των κινδύνων. Στα πρώτα ε, στρώματα, στα πρώτα επίπεδα, οι γεωργοί αναλαμβάνουν περισσότερους κινδύνους και δεν χρειάζεται μετακύληση του κινδύνου ή αν χρειάζεται μεταφορά του κινδύνου, η ανάγκη κινδυνου η αναγκη προσφυγή σε μια διαχείριση των χρήσεων, δηλαδή στην ad hoc, ε, στις ad hoc ενισχύσεις, που είναι η κορυφή της πυραμίδας, είναι λιγότερο απαραίτητη. Και γίνεται μια συνολική αντιμετώπιση των κινδύνων. Δεδομένων όλων αυτών των στοιχείων, σε τι συμπεράσματα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στη μελέτη μας. Καταρχήν διαπιστώνουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ισχύει ένα ομοιόμορφο, ομοιογενέ πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων ή για τα μέσα διαχείριση κινδύνων. Και άρα τα κράτη-μέλη αναπτύσσουν ε, τα δικά του μοντέλα που είναι διαφορετικά μεταξύ του και διαφέρουν και ω προ τι πηγές χρηματοδότηση, και ω προ τις καλύψεις και ω προ τα μέσα γιατί προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κινδύνου και ανάγκε τη κάθε χώρα. Οπότε οποιαδήποτε δυνητική μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου ή των μέσων θα πρέπει να είναι συμβατή με τα υφιστάμενα μοντέλα που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Οι κίνδυνοι θα πρέπει να διαρθρώνονται σε επίπεδα, σε στρώματα. Γιατί δεν είναι τα διάφορα μέσα και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα διάφορα μέσα δεν είναι άσχετο με το επίπεδο κινδύνου. Αυτή λοιπόν η διαστρωμάτιση των κινδύνων επιτρέπει καλύτερη συνεργασία και συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου κλάδου. Επίσης, οποιαδήποτε στήριξη των μέσων διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να λάβει υπόψη τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, των διαφόρων στρωμάτων κινδύνων. Επίσης, έγινε μια ανάλυση των στοιχείων που είχαμε στη διάθεσή μας για τα μέσα στήριξη που χρησιμοποίησαν τα κράτη-μέλη. Κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ισχύοντα μέτρα και οι κανόνες είναι αναποτελεσματικοί για την αποτροπή ή την παρεμπόδιση των κρίσεων. Δεν υπάρχουν αρκετά προληπτικά μέτρα. Οπότε τα κονδύλια που προβλέπονται για ad hoc ενισχύσεις ε, μετά την έλευση της κρίσης ε, είναι πολύ ε, πιο υψηλά. Σε ό,τι αφορά την, κατά... την κάλυψη των κινδύνων των αγορών, εδώ έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Καταρχήν πρόκειται για ένα εργαλείο το IST ε, που χρησιμοποίησε κυρίως η Ιταλία και η Ουγγαρία και η περιοχή Καστίγια Ιλαιών στην Ισπανία. Η Ιταλία είναι η χώρα που αφιερώνει περισσότερα κονδύλια στα πλαίσια του μέσου σταθεροποίηση του εισοδήματο. Οι υπόλοιπε χώρε χρησιμοποιούν πολύ μικρότερα ποσά και μάλιστα στα πλαίσια αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα αμοιβαία κεφάλαια δυστυχώ χρησιμοποιούνται ελάχιστα, όπω είδαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κράτη-μέλη. και στην επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η κάλυψη των κινδύνων των αγορών θα πρέπει προαιρετικά να καλύπτεται από ασφαλίσεις. Γιατί ασφάλειες, ασφαλίσεις είναι τα μέσα που χρησιμοποιούν κατεξοχήν οι γεωργοί στα διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, μπορούν να εφαρμοστούν ασφαλίσεις ε, εισοδήματος ε, ή εσόδων. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει τεχνικές μελέτες, μέσα για την εκτίμηση των ζημιών, ανάπτυξη αξιόπιστων δικτών εισοδημάτων ή εσόδων, δημιουργία βάσεως, βάσεων δεδομένων και αναζήτηση των συμπληρωματικών στοιχείων με τα υφιστάμενα συστήματα. Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο που θα πρέπει να γίνει. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η αντασφάλιση, η ανάγκη αντασφάλισης και σε μια κουλτούρα διαχείρισης ε, των κινδύνων των αγορών. Είναι σημαντική αυτή η δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να προσδιορίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο κάποια πλαίσια είτε συνασφάλισης είτε αντασφάλισης και μάλιστα σε συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Δεδομένου όλων αυτών των συμπερασμάτων τη μελέτη, σε τι συστάσει θα μπορούσαμε να καταλήξουμε. Η πρώτη σύσταση είναι ότι πιστεύουμε πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ε, δημιουργήσει μια δέσμη κοινών μέτρων για να ρυθμίσει ε, τα μέσα διαχείρισης κινδύνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Γεωργικών Αγορών ε, θα επέτρεπε τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την αυτόματη ενεργοποίηση και τη διαφανή ενεργοποίηση μέσων διαχείρισης των κρίσεων. Άλλο σημαντικό σημείο θα ήταν η ανάγκη οι οργανώσει των παραγωγών και οι ενώσει οργανώσεων παραγωγών να μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα για την προσαρμογή ε, της παραγωγής σε ποσότητα και ποιότητα, προκειμένου η διαχείριση των κρίσεων είναι αποτελεσματική και μάλιστα σε προληπτικό επίπεδο, πριν ε, εξελιχθεί πλήρως. Φυσικά με σεβασμό των συνθήκων και όρων του ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που μειώνονται οι βασικές ενισχύσεις, τα μέσα διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την δυνατότητα χορήγησης κουπονιών με αντίστοιχη, σε αντίστοιχο ποσό από αυτό, σε αυτό τη μείωση των βασικών ενισχύσεων, ώστε με αυτά τα κουπόνια να μπορούν οι γεωργοί να καλύπτουν κάποια μέσα διαχειρίσης των κινδύνων. Το ισχύον αποθεματικό της κρίσης αποδείχθηκε, αποδείχθηκε αναποτελεσματικό δεδομένο των κονδυλίων που αφιερώνουν τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να προγραμματιστεί εκτός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για να είναι πιο αποτελεσματικό αυτό το αποθεματικό των κρίσεων. Επίσης, η εφαρμογή μέσων διαχείρισης των κρίσεων προϋποθέτει μια ενίσχυση ικανοτήτων και προγράμματα κατάρτισης που θα μπορούσαν να περιληφθούν ειδικά στα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου. Και τελευταία σύσταση, όλα τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται με ολοκληρωμένο τρόπο στο ίδιο πλαίσιο, είτε στον πρώτο πυλώνα, είτε στο δεύτερο πυλώνα, είτε σε ένα ειδικό πυλώνα διαχείριση των αγορών πάντως ε, με συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο στην κοινή γεωργική πολιτική, λαμβάνοντα υπόψη τα διάφορα επίπεδα κινδύνου και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Αυτά σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μπαρδαχή. Όπως σας είπα και στην αρχή, θα ακούσουμε τις ερωτήσεις και τα σχόλια των Ευρωβουλευτών. Οπότε όποιος θέλει το λόγο παρακαλώ να το δηλώσει. Πρώτη κυρία Πετήρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Μπαρδαχή για την παρουσίαση της μελέτης που μας έκανε. Θα ήθελα με συγκεκριμένα παραδείγματα να μας κάνετε συστάσεις ε, για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις κρίσεις στη Γεωργία. Γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο ε, η γεωργία μας στα κράτη-μέλη είναι εκτεθειμένη σε πολλούς και διάφορους κινδύνους. Ε, πολύ συχνά πλήττονται από θεομηνίες. Και μάλιστα στην κεντρική Ευρώπη, στη Σλοβενία, την Κροατία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία είχαμε τέτοια προβλήματα φοβερών πλημμυρών αργότερα και η Γαλλία επλήγει και από παγετό και χαλάζια και οι ζημίες έχουν απολογιστεί σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Φυσικά τα κρατημέλη δεν μπορούν από μόνα τους να καλύψουν τόσο υπέρογγες ε, ζημίες, ούτε και ασφαλίσεις μπορούν να καλύψουν τις ζημίες των γεωργών και ζητήσαμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, στο συγκεκριμένο αυτό παράδειγμα, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς η διαχείριση τον κινδύνο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ή να βοηθήσει τους γεωργούς σε τόσο σοβαρές θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Θα ήταν μια λύση, για παράδειγμα, η πρικοδότηση με περισσότερα κονδύλια του αποθεματικού της κρίσης. Πιστεύετε ότι μια αύξηση του αποθεματικού της κρίσης ε, είναι σκόπιμη χωρίς όμως να επηρεάσουμε το γεωρικό προϋπολογισμό. Από πού θα μπορούσαμε να επηρεασουμε το γεωργικο προπολογισμό. επιπλέον χρηματοδοτικά μέσα για το αποθεματικό της κρίσης και πώς θα μπορούσαμε είτε να, προβλέψουμε, να προλάβουμε είτε να βλύνουμε την, τις, τις κρίσεις που πλήττουν τους Γιώργους, όπως στην περίπτωση θεομηνιών και φυσικών καταστροφών, για παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριε Χέιτεμα. Yes, thank you very much, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και σας κυρία μου για την παρουσίαση του θέματος. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Πρώτη, Από αυτά τα εργαλεία αντιμετώπισης κινδύνων ή διαχείρισης κινδύνων δεν γίνεται μεγάλη χρήση ακόμη. Γιατί εφόσον προσφέρει περισσότερο χώρο για τον ίδιο τον τομέα, για την ανάληψη των πρωτοβουλειών αυτών, που είναι πιο κατάλληλες για την αντιμετώπιση των κινδύνων και πιο κατάλληλες και για τη χρήση από τις χώρες μέλη. Γι' αυτό ρωτώ, θεωρείτε ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χώρο στην νομοθεσία και για τις ε, πρωτοβουλίες αυτές. Δεύτερο, δεύτερη ερώτηση. Βλέπετε ότι και στο δεύτερο πυλώνα δεν γίνεται μεγάλη χρήση αυτών των φωτοβουλίων. Και αν δεν κάνω λάθο, δεν είναι στοχευμένο ο δεύτερο πυλώνα εδώ. Πρόκειται να γίνει ε, στόχευση, δηλαδή διάθεση χρημάτων και στο δεύτερο πυλώνα για αυτά τα εργαλεία διαχείριση του κινδύνου. Και τέλο το πράσινο καλάθι του 30% του ΠΟΕ. Είναι άραγε απολύτως αναγκαίο να συμμορφωθούμε με το 30%. Ακούω από πολλού γεωργού ότι θεωρούν το 30% που καλούνται να δαπανίσουν εξιδίων πόρων ε, το κρίνουν υπερβολικό. Και είναι αναγκαίο να είναι και μέσα στο πράσινο καλάθι. Μπορούν να είναι και στο κίτρινο ή μόνο σε αυτό. Πορτοκαλί, πορτοκαλί καλά. Ε, η κυρία Σάιερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ε, παρουσίαση, πραγματικά με εντυπωσίασε. Θα ήθελα, ε, μας από το εξής, πέρσι στην Ολλανδία σημειώθηκε ε, μεγάλη ζημία από τροκτικά. Γι' αυτό ρωτώ, τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη. Ρώτησα και στην Κομισιόν και μου είπαν ακριβώ αυτό που είπατε και εσεί τώρα. Από τον δεύτερο πυλώνα δηλαδή τη αναπτύξεω τη υπαίθρου, ότι εκεί υπάρχει κάποια δυνατότητα. Φάνηκε όμω καθαρά ότι ο δεύτερο πυλώνα χρησιμοποιείται για άλλου σκοπού. Και εγώ εξεπλάγει για, ε, από όλε αυτέ τι δυνατότητε που υπάρχουν ε, από αυτόν τον πυλώνα. Δηλαδή, για παράδειγμα, για την προστασία τη φύσεω. Είναι δυνατόν αυτό. Ε, μπορούμε να το μετατοπίσουμε αυτό στις, ε, ε, χωρισμένη, Όταν στην Φρισλανδία έκανα τη σχετική πρόταση μου είπαν ότι δεν το γνωρίζουν αυτό. Χρειάζεται λοιπόν πολύ περισσότερη εργασία διαφωτίσεως εν τέλει για τι δυνατότητε που δίδονται. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Σένρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες για τη μελέτη που μας παρουσίασαν και να σχολιάσω το ζήτημα του κινδύνου των αγορών. Είναι μια συζήτηση που έχουμε τακτικά στη συνεδρίασή μας. Και μιλάμε συνήθως για εκούσια μέτρα, προαιρετικά. Το ίδιο λέει και οι μελέτη μέτρα προσαρμογής της προσφοράς. Μιλήσατε για ποσότητα και ποιότητα. Και κάτι άλλο που επισημάνατε είναι ότι υπάρχει δυνατότητα μείωσης των ενισχύσεων για να διευρυνθούν τα κονδύλια του Ταμείου. Δεν εξετάσετε καθόλου στη μελέτη σας η δυνατότητα αυτά μέτρα προσαρμογής, προσφοράς και ζήτησης να γίνεται μέσω δημόσιων πολιτικών που θα υποχρεώνουν τους γεωργούς στην τήρηση αυτών των μέτρων. Θα πρόκειται δηλαδή για υποχρεωτικά μέτρα και η μείωση της, ε, των πληρωμών, η μείωση των ενισχύσεων δεν θα επηρεάσει αρνητικά το ήδη συρρυκνωμένο εισόδημα των γεωργών. Γιατί οι ενισχύσεις αυτές θεσπίστηκαν γιατί είχαν ε, εφαρμοστεί πολιτικές που έχουν αρνητικές συνέπειες και ρίχνουν όλο και περισσότερο τις τιμές. Και αυτές οι ε, βασικές ενισχύσεις ήταν μια μικρή αποζημίωση ε, για την επιβίωση των γεωργών. Αν τώρα προβλέπεται μείωση, περαιτέρω μείωση, αυτών των ενισχύσεων για να αντιμετωπιστεί η εγκατάλειψη της δημόσιας πολιτικής ε, που θα οδηγήσει σε απόλυτη κατάρρευση του γεωργικού εισοδήματος, ότι τι να πω. θα εκμηδενιστεί τελείως το γεωργικό εισόδημα. Φανταστείτε να λέγαμε σε έναν υπάλληλο ότι όχι μόνο θα υποστεί μείωση μισθού, αλλά εκτός της μείωσης μισθού θα του αφαιρεθεί από το μισθό και μία ποσότητα για να χρηματοδοτηθεί ένα ταμείο που δεν ξέρουμε γιατί θα ε, χρησιμοποιούνταν ή σε τι θα εξυπηρετούσε. Γιατί κάτι τέτοιο μου λέτε για τους Γιώργους τώρα εξετάσετε στη μελέτη την πιθανότητα υποχρεωτικών μέτρων και δημόσιων πολιτικών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την παρουσίαση που μόλις ακούσαμε. Όπως είπε η Δόκτωρ, η Ιταλία, η χώρα μου, έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα για τα εργαλεία σταθεροποίηση, τα IST. Ακόμα βρισκόμαστε στη φάση βεβαίω του προγραμματισμού, γιατί θα αρχίσει να ισχύει από το Γενάρη τη Ερχόμενη χρονιά. Και οι ερωτήση που θέλω να σα κάνω έχει σχέση ακριβώ με αυτό. Στην Ιταλία το σχετικό ταμείο μάλλον, τα κονδύλια θα αρχίσουν να ταμιεύονται και να χρησιμοποιούνται από το Γενάρη. Τι θα γίνει όμως αν το Ταμείο έχει διαρκείς απώλειες για πάνω από ένα χρόνο. Τι κίνδυνος υπάρχει το Ταμείο αυτό να πτωχεύσει τι μηχανισμός μπορεί να διασφαλίσει την ε, εξακολούθηση λειτουργίας των ε, εργαλείων αυτών σταθεροποίησης των ΑΕΣΤΗ. Και αυτό με οδηγεί και σε μια άλλη σκέψη. Δεν υπάρχει κίνδυνο επανεθνικοποίηση των διάφορων πολιτικών. Μήπω είναι πιο σκόπιμο να γίνει ένα ευρωπαϊκό ταμείο και τα κράτη να εφαρμόζουν τα δικά τους εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματο, διότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη κατακαιρματισμένη έτσι. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω για την παρουσίαση και έχω μια σύντομη ερώτηση για τη διαχείριση κινδύνου. Έχει να κάνει με την κοινοτομία. Καινοτομία στον τομέα της γεωργίας. Διότι και εμείς γνωρίσαμε παγετώνες φέτος, παγετούς μάλλον, και η παραγωγή ίνου καταστράφηκε. Τα αμπέλια μας δεν τα κατάφεραν. Αν υπήρχαν ειδικέ τεχνικέ, με ειδικέ τεχνολογικέ λύσει, μπορεί και να τα σώζαμε. Οι γεωργοί μου είπαν ότι στη γεωργία, προφανώ, η καινοτομία είναι κάτι το υπέροχο. Αλλά δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Δεν έχουν πρόσβαση. Οπότε, δεν νομίζω ότι το θέμα της καινοτομίας δεν πρέπει να αποτελεί μέρος της διαχείρισης κινδύνου. Κάτι πρέπει να γίνει για να έχουν πρόσβαση πιο εύκολα οι Γεωργοί. Σα ρωτώ λοιπόν, εάν ξέρετε τι συγκεκριμένη εργαλεία θα μπορούσαν να δίδουν κίνητρα στου Γεωργού για να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ακριβώ περισσότερο τι καινοτόμε λύσει που προτείνονται. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια έρευνα και ανάπτυξη στα πλαίσια τη καινοτομία και δεύτερον, θα πρέπει να τα γνωρίζουν οι Γεωργοί για να μπορούν και να τα χρησιμοποιήσουν. Νομίζω ότι με αυτήν την έννοια, η Επιτροπή θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους γεωργούς να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον για την κοινοτομία. Αν και δεν νομίζω ότι η εξάντε ε, κοινοτομία θα μπορούσε να είναι μέρο αυτού του συστήματο διαχείριση των κινδύνων. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Αντριέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε για τη μελέτη που εκπονήσατε. Είμαι μεταξύ αυτών που συμμερίζουμε τις παρατηρήσεις σας για την προσαρμογή των εργαλείων που χρειάζεται. Και όπως είπε ο συνάδελφος Δεκάστρε, κοιτάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή τον κίνδυνο επανεθνικοποίησης των διαφορών πολιτικών, ιδίως για αυτόν τον τομέα, κάτι που θα ήταν πραγματικά επιζήμιο αν συνέβαινε. Επίσης, τα εργαλεία που θα υλοποιήσουμε, που μπορεί να υλοποιήσουμε, πρέπει να δούμε αν είναι σκόπιμα και να κοιτάξουμε για παράδειγμα την αγορά του γάλακτος. Μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση κατεπίγουσα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Στο βαθμό που το. Έτσι καλώ το Συμβούλιο θα συνέλθει την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα μπορέσει να δει πώ έχουν οι εξελίξει ω τη στιγμή εκείνη. Πάντω, ω σήμερα βλέπουμε ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για την διαχείριση του κινδύνου είναι να αντιμετωπίσουμε κυρίως τη μεγάλο αριθμό πτωχεύσεων που είχαμε πρόσφατα στη δική μου την περιοχή. Ε, μεγάλη γαλακτοπαραγωγή, ε, πολύ μάλλον γαλακτοπαραγωγή στις ορεινές περιοχές, στο πιεμό, δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να πτωχεύσουν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε λιγάκι τι γίνεται και στην πράξη, στις διάφορες περιφερειές και επαρχίες μας. Εάν ο παραγωγός αποφασίσει να μειώσει την παραγωγή του αυθορμήτως και να ε, μειώσει και την ποσότητα γάλακτος που διαθέτει στην αγορά, θα μπορούσε η Επιτροπή να το λάβει αυτό υπόψη της και να ανταποκριθεί ένα λόγος. Αλλά όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα στη σχετική συνάντηση, πρέπει να υπάρξουν ε, μέτρα δραστικά. Θα πρέπει να υπάρξουν και τα απαραίτητα μέσα και ε, τα κονδύλια να ανταποκρίνονται και στις ανάγκες της προσφοράς Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε. Θα πρέπει το Συμβούλιο του Ιουνίου ή το πλέον αργότερο τον Ιούλιο να δώσει πια μια απάντηση σε όλα αυτά τα θέματα, διότι θα είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ κύριε Σροπέ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, Ισαβέλα Μπαρταζή για την παρουσίαση του θέματος που βρίσκω ότι είναι πραγματικά σημαντικό και πρέπει όντως να εγκύψουμε περισσότερο στα συμπεράσματα της μελέτης, να αναλύσουμε τα εργαλεία που ισχύουν και βεβαίως και αυτά που θα χρησιμοποιήσουν και στο μέλλον γιατί είναι και διαφορετικός ο χρόνος που χρησιμοποιούνται τα διάφορα ε, εργαλεία των εισαγωγικών. Πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται τώρα και να είμαστε και αισιόδοξοι για το μέλλον. Όλοι βεβαίως θέλουμε να διαμορφωθεί καλύτερα το μέλλον. Όλοι θέλουμε οι νέοι να εισέλθουν ε, στην γεωργία. Βεβαίως οι συνθήκες ποικίλουν και ε, δεν εξαρτώνται όλα από τη συγκεκριμένη χώρα μέλος. Υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες, ε, ισχύουν διαφορετικά φορολογικά συστήματα διαφορετική δασμή Για παράδειγμα στην Λιθουανία η κυβέρνησή μας ε, επιβάλλει τέλος καταναλώσεως στο καύσιμο ντίζελ το οποίο οδήγησε σε αύξηση των δαπανών των ε, παραγωγών όπου δεν ε, δόθηκε καμιά αποζημίωση. Βεβαίως το εισόδημα του γεωργού εξαρτάται από τις τιμές που πληρώνει για τα διάφορα προϊόντα που χρησιμοποιεί και από τις τιμές που εισπράττει πουλώντας στην αγορά τα προϊόντα που παράγει. Ε, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Και όπως εξήγησα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Μάλιστα, ε, ορισμένες φορές η αστάθεια των τιμών είναι πολύ έντονη. Και οι τιμές μπορούν να ανέβουν ή να κατέβουν μέχρι και 200%. η αγοραστική δύναμη των γεωργών είναι τελικό το θύμα. Πρέπει να ενισχύσουμε τους γεωργούς ώστε να έχουν και ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη σωστή ενημέρωση των γεωργών για τους διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα η αστάθεια των τιμών, ώστε τελικά να μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερο εισόδημα στην Λιθουανία αλλά και σε άλλες χώρες. Ο, το ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται με τη γεωργία είναι πολύ περιορισμένο. Και σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο, είναι πολύ δύσκολο να εισαχθεί το στοιχείο του καταμερισμού του κινδύνου. Οι γεωργοί απλώς προσπαθούν να επιβιώσουν. Και βεβαίως οι υπόλοιποι στην αλυσίδα της διατροφής το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να μειώσουν το κόστος των προϊόντων που αγοράζουν. Χρειάζεται λοιπόν να εισαγάγουμε μέτρα τα οποία να είναι αποτελεσματικά, να είναι εναρμονισμένα στο ευρωπαϊκό επίπεδο διότι στο εθνικό επίπεδο τα μέτρα εισάγονται με υπερβολικά αργό ρυθμό και αυτό οδηγεί σε πολλές πτωχεύσεις εκμεταλλεύσεων. Πέρσι στην Λιθουανία χρειάστηκε τόσος χρόνος για τις διαβουλεύσεις σχετικά με ορισμένα μέτρα που τελικά η αξία τους στην πράξη, η αξία των νομοθετικών αυτών μέτρων στην πράξη, όταν τελικώς τα μέτρα αυτά επιβλήθηκαν ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Άρα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύτερα, παρά να προσπαθούμε να τα αντιμετωπίζουμε ατομικά εντό εισαγωγικών στο επίπεδο της κάθε χώρας μέλους. Γιατί αλλιώς θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα μείνουν πλέον εκμεταλλεύσεις στον αγροτικό τομέα. Για παράδειγμα, το ε, σύνολο των αγελάδων στη Λιθουανία έχει ήδη μειωθεί κατά 20% πολλοί εγκαταλείπουν την κτηνοτροφία. Χρειάζεται λοιπόν να τους εξασφαλίσουμε εισόδημα πριν να πτωχεύσουν όλοι αυτοί. Ε, εσείς κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της μελέτης. Είμαι και ιδιαίτερο ικανοποιημένη που μας δόθηκαν συγκεκριμένα ε, λεπτομερή νούμερα. Έχουμε τώρα το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2013 έως 20 και λάβαμε τώρα και τη σχετική τεκμηρίωση από την κυρία Μπαρδαχή και βλέπουμε ότι λίγες χώρες χρησιμοποιούν τις δυνατότητες αυτές. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει τα αίτια και να σκεφτεί αν όντως μπορούμε να βρούμε μεταξύ 28 χωρών μελών μια βάση ώστε να εφαρμόσουμε ε, ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Παρόλο που είναι σαφές για μένα ότι ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα στις διάφορες χώρες μέλη οδηγούν στο να μην έχουμε μια πραγματική κοινή αγροτική πολιτική. Κάθε χώρα μέλος δρά για λογαριασμό της. Θεωρώ σωστό να δημιουργηθεί ένα ταμείο κρίσεως ξεχωριστά, εκτός δηλαδή του δημοσιονομικού πλαισίου για να μπορούμε να αντιδρούμε τάχιστα και να προσφέρουμε πραγματική βοήθεια. Είναι σαφές επίσης ότι και εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας θα χρειαστεί να συζητήσουμε αρκετά εντατικά εάν όντω θέλουμε οι άμεσες πληρωμές όντω να μειωθούν, να μειωθούν σημαντικά και τα χρήματα να πηγαίνουν σε ένα ταμείο ασφαλίσεως. Διότι ένα είναι σαφές, οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις που όλοι εδώ επιθυμούμε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε, οι μικρές αυτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις εξαρτώνται περισσότερο από τις άλλες, από τις άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα. Και νομίζω ότι έχει έρθει όντως η ώρα να εξετάσουμε τους μηχανισμούς που μπορούν να τις εξασφαλίσουν τις μικρές αυτές επιχείρησεις, τις μικρές εκμεταλλεύσεις. ώστε να αντιμετωπιστούν και οι τρέχουσες κρίσεις και οι μελλοντικές. Άλλωστε, στις ΗΠΑ προτείνεται ένα ενιαίο σύστημα. Ας εξετάσουμε και εμείς αν μπορούμε κάτι τέτοιο να κάνουμε εδώ μεταξύ των 28 χωρών μελών της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σουλουαζό. Oui, merci, Ευχαριστώ πρόεδρε. Το γνωρίζετε και ο ίδιος η Γεωργή σήμερα δεν ζητούν απλώς να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω θέλουν εργαλεία πρόληψης των κινδύνων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει δημόσια παρέμβαση. Όμω αυτή τη στιγμή με την ε, σύναψη των συμβάσεων σε προηγούμενε φάσει ε, όλα έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Η κρατική στήριξη σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων έχει αντικατασταθεί από διαχείριση των κινδύνων μέσω των ασφαλιστικών ή των αντασφαλιστικών ταμείων με την υποχρεωτική συνδρομή. Έτσι στη Γαλλία λόγου χάρη το σύστημα αυτό των ιδιωτικών εισφαλιστικών έχει υποκαταστήσει το Εθνικό Ταμείο ε, της ε, ε, αντιμετώπισης των θεομηνιών για τον τομέα των ενοπληματοδών, λόγου χάρη. Αυτό που ήταν μια πραγματική δέσμευση του κράτους απέναντι στους ίδιους τους γεωργούς. Ε, σε σχέση λοιπόν με τι διατάξει διαχείριση των ε, ταμείων αυτών και επειδή μα ενδιαφέρουν και οι περιβαλλοντικοί και οι υγειονομικοί ε, κανόνες κανόνε και το πόσο μπορεί να αντέχουν να πληρώνουν τι συνδρομέ του οι γεωργοί που είναι ενθελούσιε ή υποχρεωτικέ και είναι ένα επιπλέον βάρο για του κτηνοτρόφου και γεωργού, αν είναι 20 ευρώ το χρόνο ετησίω είναι ένα πράγμα, όμως τελικά τα ποσά είναι τελείω διαφορετικά ανάλογα με τον εξειδικευμένο τομέα. Οι γεωργοί λοιπόν και οι κτηνοτρόφοι έχουν καμία δυνατότητα αποζημίωση μέσω των ταμείων αυτών, διότι οι όροι είναι αυστηροί και έχουν να κάνουν και με τι πρακτικέ καλλιέργειε. Και αυτό έχει να κάνει και με το πώ λειτουργεί το Ταμείο Αμεβιοποίηση των Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Κινδύνων. Δεν υπάρχουν λοιπόν άλλε στρατηγικέ πιο αποτελεσματικέ ώστε οι γεωργοί να μην είναι παραδομένοι ε, στι ασφαλιστικέ και κατ' επέκταση και στι τράπεζε και στα συμφέροντά του. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπόκοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για ένα σημαντικό κλάδο Ο κλάδο αυτό είναι πολύ σημαντικότερο τώρα από ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Είναι πολύ μεγάλη η επισφάλεια και η διακυμάνωση των τιμών στην αγορά και αυτό σημαίνει ότι οι γεωργοί θα έχουν χειρότερα προβλήματα στο μέλλον, ακριβώ λόγω των διακυμάνσεων των τιμών. Και υπάρχουν και πολλέ απρόβλεπτε φυσικέ καταστροφέ, θεομηνίε. Προσφάτω, λόγω χάρη, είχαμε παγετό στις, ε, στους οπορώνες και στους αμπελώνες μας. Και αντί να έχουμε 150 τόνους μήλα σε κομιδή, έχουμε 10 ή 15 εν τέλει. Προσωπικώς έχω πείρα από τέτοιου είδους θεομηνίες. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας, αλλά έχω και την εξής ερώτηση τι θα πρέπει να κάνουμε εδώ στην Ευρώπη για να πετύχουμε αυτό που οι Αμερικανοί φίλοι μας από τις ΗΠΑ Πολιτείες μας είπαν ότι κάνουν. 80-90% όλη ε, όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να είναι ασφαλισμένες. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν νομίζω μεγαλύτερες προσπάθειες και να κοιτάξουμε να διασφαλίσουμε ό,τι μπορεί να διασφαλιστεί Δηλαδή 10% μόνο από τους οπορώνες είχαν ασφάλεια θέτος. Όσοι εργάζονται στον τομέα του γάλακτος λόγου χάρη λένε κάτι ανάλογο, ότι χρειαζόμαστε ε, αποτελεσματικά εργαλεία και θα πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή για να υπάρχει ένα σύστημα δίκαιης αποζημίωσης και αντιστάθμισης. Θα πρέπει δηλαδή να αυξήσουμε το βάρος της χρηματοδότησης ε, αυτών των μέτρων, διότι στις ΗΠΑ 2 τρίτα ή 80% όλης της χρηματοδότησης χρησιμοποιείται ακριβώ για τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ στην Ευρώπη μόνο 1% των κονδυλίων ε, κατευθύνονται εκεί. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Η... Μήπως έχει φτάσει η ώρα για να χρησιμοποιήσουμε στο 1 τέταρτο ή 1 τρίτο τη χρηματοδότηση τη ΚΑΠ, των κονδυλίων τη ΚΑΠ για τέτοια μέτρα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε φρέσκια νέα χρηματοδότηση να φτάσει στα χέρια μα σύντομα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε εντό τη υπάρχουσα γεωργική πολιτική. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά εργαλεία και από αυτή την έννοια, με αυτόν τον τρόπο, να έχουμε ένα σταθερότερο ε, τοπίο για τι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Περισσότερα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν για τη διαχείριση των κινδύνων, ιδάλω οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι θα πτωχεύσουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Ντέ. Ευχαριστώ ε, αγαπητέ πρόεδρε. Επειδή κάποιος μίλησε για το αμερικανικό σύστημα, εγώ ξεπλάγει με τον τρόπο που παρουσίασαν το σύστημα οι Αμερικανοί δεν αφορά την κτηνοτροφία. Είναι μονάχα για τις καλλιέργειες. Εμείς έχουμε ήδη συστήματα ασφαλίσεων, για παράδειγμα κατά του χαλαζιού ή των ζημιών από καταιγίδε. Οι είναι είναι ασφαλισμενη Και η τρέχουσα γεωργική πολιτική επιτρέπει στις χώρες μέλη να χρησιμοποιήσουν κονδύλια για συστήματα ασφαλείας, αρκεί να εφαρμοστεί αυτό ότι χρειαζόμαστε κανόνες πανευρωπαϊκής εμβέλειας ε, ενάντια των θεομηνιών, αυτό είναι σαφές. Αλλά τώρα ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας, η ασφαλίσεως, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, διότι είναι πολύ διαφορετικές 28 χώρες μέλη. Δεν είναι δυνατόν να οργανωθεί κάτι τέτοιο από τις Βρυξέλλες. Θεωρείτε ότι, θεωρώ μάλλον, ότι είναι πολύ έντονο το στοιχείο της εθνικής ευθύνης, ακόμα και αν διατίθεται και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις περιπτώσεις όπου μετακινούμε στην Βαβαρία χθες, πολλοί γεωργοί μου λένε ότι το πιο σημαντικό για αυτούς είναι να δουν αλλαγές στο εθνικό φορολογικό δίκαιο, είτε για την, για την ε, κτηνοτροφία γενικότερα, είτε για τη χειροτροφία, να μπορούν να δημιουργούν αποθεματικά αφορολόγητα στα καλά έτη για να είναι ασφαλισμένοι για περίπτωση όπου κάτι δεν θα πάει καλά μια χρονιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Νταουντάμ. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτη όταν συγκρίνουμε με άλλους και ιδίως με το αμερικανικό σύστημα, είναι σαφές ότι εμείς εξακολουθούμε να ε, είμαστε θεματοφύλακες της συμφωνίας του Μαρακές. Ένα στοιχείο που νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε υπόψη. Δεύτερο στοιχείο, στην μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής, οφείλω να θυμίσω ότι το Κοινοβούλιο ήθελε να προχωρήσει περισσότερο για ορισμένα θέματα για παράδειγμα για τον ΠΟΕ και ιδίω για τα ε, φρούτα και κυπευτικά και για το κρασί. Όμως δεν έγινε τελικά αυτό. Εγώ συμφωνώ με τον Άλμπερντες που έχει εξετάσει το θέμα. Το δίκαιο, το ασφαλιστικό δίκαιο των χωρών μελών είναι τόσο διαφορετικό που θα είναι πολύ δύσκολο στις περισσότερες περιπτώσεις να εφαρμοστεί ένα κοινό σύστημα. Οφείλει κανεί να λάβει υπόψη την διπλωματικότητα αυτή. Η κοινή αγροτική πολιτική βάζει κάποιε κατευθύνσει, διαθέτει εργαλεία και εξαρτάται από την κάθε μια χώρα μετά να τα εφαρμόσει τα εργαλεία αυτά, να τα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτά σύμφωνα με το εθνικό τη δίκαιο. Όπω έχουν εξελιχθεί οι ασφαλίσει, δείχνουν μία από τι λύσει απέναντι στι κρίσει και στην αστάθεια των τιμών. Δεν μπορούμε να μείνουμε εμεί οι Ευρωπαίοι οι μοναδικοί στο περιθώριο αυτού του συστήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ολοκληρώσαμε το κατάλογο με τους ομιλητέ μας. Δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο. Δεν θα ξέρω αν ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να μιλήσει. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. No, simply... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, απλώ να πω και εγώ ότι καλωσορίζουμε τη μελέτη. Είναι χρήσιμη συνεισφορά στην τωρινή μα συζήτηση για το ποια ήταν η πρόσληψη των εργαλείων διαχείριση του κινδύνου, κυρίω για το εργαλείο σταθεροποίηση του εισοδήματο στην Ευρώπη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τι σχετικέ ενέργειε και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με του συντάκτε τη μελέτη για να ενισχύσουμε περαιτέρω την κατανόηση του γιατί η πρόσληψη και η χρήση του εργαλείου έγινε με τέτοια βραδύτητα, ώστε στο μέλλον να επιταχύνουμε την αξιοποίηση ανάλογων εργαλείων. Μπράβο σας για τη μελέτη, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά όμως, για την οποία είμαστε ανυπόμονοι και πρόθυμοι να συνεισφέρουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο σε εμπειρογνώμονές μας, στους καλεσμένους μας, για να σχολιάσουν και να απαντήσουν ε, στις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Συνεννοηθείτε εσείς ποιος ε, θα πάρει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά για να ξεκουραστούν λίγο οι διερμηνείς και Υπάρχουν ε, πολλές ερωτήσεις, τις σημειώσαμε και με μεγάλη χαρά, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, ίσως όχι τώρα, όχι αμέσως, λεπτομερώς, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ήθελα να επιμείνω σε δύο σημεία, στην ε, συνοχή και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όταν ε, καταρτήσαμε αυτή την πυραμίδα, θελήσαμε να τονίσουμε τη σημασία της συνοχής σε σχέση με τη διαφορετικότητα, την ποικιλία των πολλών φορέων και δράσεων. Το να προωθήσουμε τη διαχείριση των κινδύνων σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων θα επιτρέψει και αυτό συσχετίζεται με στοιχεία της έκθεσης Ντόντα θα επιτρέψει να εξισορροπηθεί καλύτερα όλος κλάδος διότι οι κίνδυνοι θα είναι σωστά κατανεμημένοι καθ' όλη την αλυσίδα παραγωγή. Δεν θα βαρύνουν μόνο του γεωργού. Έτσι θα υπάρχει προληπτική διαχείριση των κινδύνων. Ο κύριο Ντεκάστρο στο βιβλίο του άλλωστε τα έχει υπογραμμίσει όλα αυτά. Την ε, σημασία τη προληπτική διαχείριση κινδύνων όπω το calming market instrument θα μπορούσε να λειτουργήσει ω ένα εργαλείο ε, καταπράινση τη αγορά. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν την δημοσιονομική οργάνωση και προληπτικά και για να ωφελήσουν τις επενδύσεις. Οι γεωργοί δηλαδή μπορούν να επενδύσουν τις καλές χρονιές και να εξοικονομήσουν τις ε, χειρότερες. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης συνοχή σε επίπεδο πολιτικό. Δηλαδή σήμερα ε, μιλήσαμε για την ΚΑΠ γενικότερα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γενικώ και για την κρίση, όμω είναι περίεργο να δούμε ότι σε κάποια κράτη υπάρχουν συνδεδεμένε βοήθειε για την γάλακτοπαραγωγή και αυτή τη στιγμή ζητάμε συνδεδεμένε βοήθειε για την ε, μείωση τη παραγωγή γάλακτο. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη συνέπεια στην όλη μα προσέγγιση. Συνέπεια απαιτείται και σε επίπεδο τη δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αγαπητοί, αγαπητοί φίλοι, ε, συνάδελφοι, για να γνωρίζουμε λιγάκι πότε θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους των διακυμάνσεων. Συνέπεια, χρειάζεται και σε επίπεδο της χρήσης των άμεσων ενισχύσεων ή των εθνικών, ώστε αυτές να μπορέσουν από κοινού να δώσουν αποτελέσματα στον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα. Έχουν γίνει και προσπάθειες όπως στη στην μεταρρύθμιση που έγινε για τις τριστικέ οργανώσεις ή την οριζόντια οργάνωση των τομέων από τον πρώτο πυλώνα και την ε, οργάνωση παραγωγών στο δεύτερο. Η συνέπεια είναι για μας ε, καθοριστική σημασίας. Έχουμε ετοιμάσει διαφορετικές συστάσεις όπως για το άρθρο 122 που αρχίζει να γίνεται ε, λογικό όταν μιλάμε για προληπτική διαχείριση των κινδύνων όπως είπε και ο κύριος Νταντέν στην έκθεσή του. Δεν έμεινε βέβαια αυτή η συμβιβαστική λύση αλλά όταν ε, ξέσπασε η κρίση ζητήσαμε από τους φορείς να τα διαχειριστούν ε, προσωπικά σε ατομικό επίπεδο. Αυτό ξεπερνάει λιγάκι όσα θελήσαμε να οργανώσουμε. Είναι λιγάκι δύσκολο ο καθένα μόνο του να σβήνει μια πυρκαγιά. Ε, συνέπεια λοιπόν και δεύτερον το κοινοτικό πλαίσιο. Πολλά μπορούν να γίνουν σε επίπεδο κοινοτικού πλαισίου για να μπορέσουν ε, να υλοποιηθούν κάποια πράγματα. Δεν είμαστε βεβαίω ότι σήμερα ένα κοινοτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τόσο διαφοροποιημένη, τόσο ποικιλόμορφη, μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη απορρόφηση των κομπηλίων. Τα επίπεδα των κινδύνων είναι διαφορετικό. Θελήσαμε λοιπόν στην έκθεση αυτή να βασιστούμε σε όσα ήδη ισχύουν σήμερα και να γίνει μια πρόταση ε, όχι για να μην αλλάξει η ΠΑΚ, ούτε και για να γίνει μια ριζική επανάσταση. Υπάρχουν συστήματα σε επίπεδο κρατών που λειτουργούν και λειτουργούν καλά. Οι δυνατότητε που υπάρχουν εν μέρη αξιοποιούνται, εν μέρη θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται περισσότερο, αλλά το υπάρχον πλαίσιο α το βελτιώσουμε. Α το βελτιώσουμε αντί να ονειρευόμαστε μια ριζική μεταστροφή και να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο το κοινωτικό πλαίσιο. Γιατί αυτό μπορεί να μην επιτρέψει την απαραίτητη διαλλακτικότητα ευελιξία που χρειάζονται σημερινέ καταστάσει. Όπω είδαμε, η κατάσταση του ενό κράτου μέλου διαφέρει πολύ από άλλα και το να θέλουμε σε κοινοτικό επίπεδο με ομοιογένεια να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση τροποκυλόμορφη δεν μου φαίνεται ο πιο σκόπιμο τρόπο. Α επικεντρώσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση στι παρεμβάσει τη εκεί που μπορεί να είναι πιο ε, αποτελεσματική. Πολλά μπορούν να γίνουν. Είπαμε για τον πρώτο πυλώνα, είπαμε για τον τρίτο πυλώνα, υπάρχει και κατάρτιση. Αυτό είναι επίση σημαντικό να το τονίσουμε. Η μάθηση για του μηχανισμού που μπορεί να υπάρχουν και να μην είναι γνωστοί. Και τελευταίο στοιχείο, σε επίπεδο κρίση και διαχείριση τη κρίση Εμάς, η όλη μας λογική δεν ήταν απλώ πώ να ξεφύγουμε από την κρίση στην Ελλάδα σήμερα, αλλά πώ να σχεδιάσουμε μια νέα ΚΑΠ με ορίζοντα το 2020 και το καθεξής. Μπορούμε πολύ να μιλάμε για την τωρινή κρίση και για το τι πρέπει να γίνει τώρα, όμως η δική μας λογική, η βασική λογική είναι ότι ο προπολογισμό τη Γεωργίας πιθανώ θα δεχτεί σοβαρότατε πιέσει τα ερχόμενα χρόνια. Το ακούμε από τόσε συζητήσει. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να γίνει, αλλά είναι σημαντικό για να έχουμε έναν προπολογισμό για τη γεωργία στο ύψο ε, των φιλοδοξιών μια Γεωργία για την Ευρώπη, πρέπει να βρούμε τα καλύτερα δυνατά εργαλεία για να μεγιστοποιήσουμε το δυτικό αντίκτυπο για του παραγωγού. Γι' αυτό δεν προτείνουμε κατάργηση των βοηθειών αλλά σχεδιάζουμε το πώς θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια και να τα χρησιμοποιήσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Προφανώς, όταν υπάρχει μια κρίση, πρέπει κανείς να ε, έχει και τους κατάλληλους μηχανισμούς. Αυτό είναι όμως άλλη συζήτηση. Συνέπεια, κοινοτικό πλαίσιο, αλλά ούτε αποκλειστικότητα του κοινοτικού πλαισίου. Μπορούμε πολλά να κάνουμε σε επίπεδο κοινότητα, αλλά και πολλά... Ε, μαθαίνοντα το τι είναι, ε, λειτουργεί ω καλή πρακτική σε ένα άλλο κράτο μέλο. Ξέρω ξέρω με τι άμεσε και έμεσε βοήθειε. Θα ήθελα και εγώ να προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις στις πολυάριθμες ερωτήσεις. Πολλοί μιλήσα, μίλησαν για την θέσπιση κοινού γεωρικού ταμείου για τις γεωρικές ασφαλίσεις ε, για κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γεωργία. Είναι λογική ιδέα, αλλά είναι πολύ ανομοιόμορφη οι κίνδυνοι που υπάρχουν στην Ευρώπη μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, μεταξύ κτηνοτροφίας και γεωργίας. Και κυρίως, αν συστήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο και αν γίνει μια αμοιβεοποίηση των γεωργικών, αγροτικών κίνδυνων στην Ευρώπη, κάτι τέτοιο ε, θα απαιτήσει μια δημοσιονομική ανακατανομή μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που είναι πολύ περίπλοκο και θα προσκρούσει σε μεγάλα εμπόδια στο Συμβούλιο. Είμαι 100% βέβαιο αυτό. Φανταστείτε αν θα πρέπει να γίνει ανακατανομή. Γιατί δεν αντιμετωπίζουν όλε οι χώρε του ίδιου κινδύνου και η αμοιβεοποίηση προϋποθέτει ανακατανομή του προϋπολογισμού. Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα είναι αυτές των ε, λογαριασμών ε, αποταμίευσης. Γιατί υπάρχουν περίοδοι παχιών και ισχνών αγελάδων, βάζουμε κάτι στην άκρη στις παχές αγελάδες για να αντιμετωπίσουμε τις ισχνές. Αυτό είναι λογικό στη θεωρία, στην πράξη όμως είναι πολύ δυσεφάρμοστο. Γιατί οι Γεωργοί, για παράδειγμα, πρέπει να έχουν αυτή την κουλτούρα της ε, οικονομίας εξοικονόμησης, κάτι που δεν ισχύει. Επίσης, ο βαθμός ενημέρωσης ε, και η διαχείριση που είναι τόσο περίπλοκη και επίσης ε, τι γίνεται με την αμοιβαιοποίηση και σε περίπτωση πτώχευσης τι γίνεται. Επίσης, το πρόβλημα της φορολογίας ε, γιατί πολύ διαφορετικά αντιμετωπίζονται στη φορολογία οι ε, λογαριασμοί ταμιαστήριου. Και όταν είναι ευνοϊκό το φορολογικό καθεστώς, ουσιαστικά ε, ενισχύεται η προσφυγή σε αυτό το μέσο. Και παραλαμβάνω, και επειδή οι φορολογίες αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους λογαριασμούς ταμιαστήριου, ε, θα είναι διαφορετική θέση στην οποία θα βρεθούν οι Γεωργοί προσφεύγουν σε αυτό το μέσο. Επίσης, οι μηχανισμοί διαχείρισης ε, κρίσεων ε, και κινδύνων δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, δεν διαδραματίζουν σωστά το ρόλο τους. Ούτε αποτελεσματικοί είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ούτε υπάρχουν σαφείς κανόνες για το πότε ενεργοποιούνται αυτοί οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων ή ενεργοποιείται το αποθεματικό κρίσης. Και αυτή η αυθαιρεσία που υπάρχει είναι πολύ επικίνδυνη. Χρειαζόμαστε σαφείς και διαφανείς επικινδυνη χρειαζομαστε σαφεις και διαφανεί κανόνε για το τι εστί κρίση, πότε ε, λαμβάνει η χώρα. Θα πρέπει να ορίσουμε τι εστί κρίση και τότε αυτόματα να ενεργοποιείται ο μηχανισμό διαχείριση των κρίσεων. Δεν μπορούμε αυθαίρετα να χαρακτηρίζουμε κάτι κρίση ή ε, μια κατάσταση ω κρίσιμη και άλλη όχι. Πρέπει να έχουμε σαφείς δείκτες, ξεκάθαρους κανόνες ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός διαχείρισης των κρίσεων, να αποφεύγεται οποιαδήποτε αυθαίρετη ενέργεια. Επίση, σε περίπτωση αποθεματικού κρίσεων θα πρέπει να είναι εκτό ε, του προπολογισμού. Γιατί αν ε, περιληφθεί στον προπολογισμό όπω ισχύει τώρα, θα έχουμε λογικά πολλέ δυσκολίε με το αποθεματικό κρίσεων. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε είναι τα προβλήματα του γαλακτοκομικού τομέα. Ένα από τα θέματα που επισημάναμε είναι ότι ε, σε τομείς που υπάρχουν παραγωγοί, οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις παραγωγών, μπορούν αυτές οι οργανώσεις να παίξουν ρόλο για να αποφύγουν την κατάρρευση των τιμών ή να την αναχαιτήσουν κάπως ή να την επιβραδύνουν. Βέβαια, το θέμα αυτό προσκρούει μερικές φορές στους κανόνες ανταγωνισμού. Υπάρχει μερικές φορές αντίφαση και το ζήτημα δεν έχει επιλύθει. Θα πρέπει πιο ενδελεχώς να εξετάσουμε ε, σε ποιο μέτρο ε, μια ενέργεια του, των οργανώσεων παραγωγών ε, δεν αντιβαίνει με τους κανόνες ανταγωνισμού. Θα πρέπει να γίνει αυτή η διευκρίνηση που είναι απολύτως απαραίτητη. Ένα άλλο σημαντικό θέμα. Η διαχείριση των κινδύνων και τα μέσα διαχείρισης κινδύνων δεν ε, έχουν σκοπό την διάσωση ενός τομέα από μια διαρθρωτική κρίση. Αν η τάση ε, των τιμών είναι ευθύνουσα επί σειρά ετών, το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό, οπότε δεν θα επιληθεί με ένα μέσο διαχείρισης κινδύνου, γιατί δεν είναι θέμα κινδύνου, αλλά διαρθρωτικής κρίση του κλάδου. Άρα χρειάζεται αναδιάρθρωση στο κλάδο. Η διαχείριση της κρίση έχει νόημα όταν ε, μια χρονιά έχουμε μείωση τιμών και άλλη όχι. Όταν έχουμε σταδιακά και συστηματικά μείωση των τιμών, το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό και εμπίπτει στη διαχείριση με μέσα διαχείριση κρίσεων. Εμεί προτείνουμε κάποιε ενδιαφέρουσε ιδέε. Για παράδειγμα, την ίδρυση παρατηρητηρίου τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταλήξουμε σε κάποιους αυτόματους δείκτες ενεργοποίησης του μηχανισμού αντιμετώπισης των κρίσεων. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μηχανισμούς, ενημέρωση, βάση δεδομένων και παρατηρητήριο τιμών. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη δουλειά και επεξεργασία όλων αυτών των προτάσεων. Και τέλος, θα ήταν σημαντικό στο Ταμείο, μία από τις προτάσεις μας που θα μπορούσε να μελετηθεί εκτενέστερα και διεξοδικότερο. Ένα από τα μέσα που δεν εφαρμόστηκε στη μεταρρύθμιση ΚΑΠΑ 2014-2020 στο δεύτερο πυλώνα είναι το θέμα των ασφαλίσεων. Ασφαλή εσόδων ή εισοδήματος. Αναφέρθηκε το θέμα των αμοιβαίων κεφαλαίων για τις εισοδίες. Ε, εφαρμόστηκαν ε, ε, μηχανισμοί λογαριασμών ταμιευτηρίου. Ακόμη και ο μηχανισμός σταθεροποίησης γεωργικού εισοδήματος το IST. Ένα από τα μέσα αυτά είναι και τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ε, λογαριασμοί του διευθυντήριου, αλλά όχι και οι ασφαλίσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε ένα νέο μηχανισμό που θα ήταν η ασφάλεια εσόδων ή εισοδημάτων που θα συμπληρώνει τις υπάρχουσες ασφαλίσεις των αποδόσεων των συγκομιδών. Νομίζω ότι αυτό το θέμα της ασφαλής εισοδήματος ή εσόδων θα ήταν ένα συμπληρωματικό μέσο πολύ χρήσιμο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, συμπληρωματικό προς τις ασφαλείς εισοδίας. Η ε, κυρία Παρταχή. θα ήθελα πρώτα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση, γιατί οι συνάδελφοι με κάλυψαν σχεδόν πλήρω. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποιες προτάσεις που έγιναν ε, για την μείωση των ενισχύσεων. Τη μείωση ενισχύσεων, των βασικών ενισχύσεων προς τους γεωργούς. Εμείς δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Απλώς ε, είπαμε ότι υπάρχει δυνατότητα μείωση της βασικής ενίσχυσης για τους μεγάλους παραγωγούς, όχι για τους μικρούς παραγωγούς. Αυτοί εκπίπτουν από την πρόταση. Οι περισσότεροι άλλωστε παραγωγή είναι μικροπαραγωγή. Αυτό είναι η βασική ενίσχυση, δεν επηρεάζεται, μένει άθικτη. Αλλά λέμε, ε, είναι δυνατό ένα τμήμα της βασικής ενίσχυσης των μεγάλων παραγωγών να ε, αφιερωθεί στα μέσα διαχείρισης κινδύνων από τους ίδιους τους παραγωγούς. Έτσι θα δίναμε κίνητρα στις μεγαλύτερες ιερικές εκμεταλλεύσεις που είναι πιο προσανατολισμένες στις αγορές να εφοδιαστούν με νέους μηχανισμούς ε, ασφαλίσεων και μεταφοράς κινδύνων και κάλυψης ε, κινδύνων αγορών. Επίσης, αναφερθήκαμε στους κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου και στην πιθανότητα να στηριχθούν κάποια μέσα για καλύψεις ε, ε, όχι σοβαρών ζημιών και κινδύνων, δηλαδή ζημιών και κινδύνων λιγότερο, χαμηλότερων του 30%. Δεν πρέπει να να μετατραπούμε ως θεματοφύλακες της Σύμφωνίας του Μαρακές, όπως αναφέρθηκε. Απλώς ε, λέμε να στηρίξουμε κάποια μέσα ασφάλισης για μη σοβαρέ ζημίες, για ζημίες που είναι λιγότερε των 30%. Τώρα ε, για ζημίες, άνω των 30% είναι τόσο καταστροφικές και ολέθριες ε, που χρειάζεται μια άλλη ε, αντιμετώπιση. Βέβαια και εδώ υπάρχει ανομιμορφία μεταξύ των διαφόρων τομέων. Πάντως Πιστεύουμε ότι η ΚΑΠ δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα μέσα του πράσινου κουτιού. Υπάρχει περιθώριο ώστε να στηριχθούν και κάποια μέτρα του πορτοκαλί κουτιού. και να στηριχθούν ασφαλίσεις για σοβαρές που δεν είναι τόσο σοβαρές, δηλαδή δεν φτάνουν στο 30%. Αυτά, ευχαριστώ. Βέβαια, ανακύπτει το ερώτημα πότε ξεσπάει η κρίση, πότε θεωρούμε ότι η κρίση. Με τι κριτήρια θα χαρακτηρίσουμε μια κατάσταση ως κρίση. Τι σημαίνει κρίση. Πότε θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα αναχέτησης της κρίσης ή πρόληψης της κρίσης. Και η πρόληψη σίγουρα είναι λιγότερο δαπανηρή όσο πιο γρήγορα αντιδράσουμε και αποτρέψουμε την κρίση, τόσο λιγότερα κονδύλια θα χρειαστούμε μετά για να την μετριάσουμε. Και έτσι θα αποτρέψουμε και την αστάθεια, γιατί εδώ η αστάθεια είναι το πρόβλημα και η ανασφάλεια όταν ε, σκεφτεί μια κρίση. Αυτό το θέμα του τι αντιλαμβανόμαστε ως κρίση είναι πολύ σημαντικό και πώς θα χαρακτηρίσουμε την κρίση. Η δική μας Επιτροπή διαφορετικά αντιδρά. Λέει, λέμε πάντα, όχι, ακόμη δεν έχουμε κρίση. Και όταν ε, φτάνει η κρίση και μας χτυπάει, λέμε, α, βλέπουμε ήδη το φως στην άκρη του τούνελ. Αλλά δεν είναι έτσι πάντα τα πράγματα. Για παράδειγμα, είδαμε τι έγινε με την γαλακτοκομική κρίση, την κρίση στο γαλακτοκομικό κλάδο. Θυμάστε την Επιτροποφή Φίσερ Το τράβηξε, το τράβηξε, καθυστέρησε μέχρι να εγκρίνει τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, με αποτέλεσμα ε, οι δαπάνες είναι πολύ μεγαλύτερες. Και χρειάστηκε κάποια αναδιάρθρωση τελικά. Και σίγουρα η αναδιάρθρωση θα οδηγούσε σε παραπλησμό πολλών γαλακτοπαραγωγών. Και γι' αυτό και η αναδιάρθρωση σε πρώτερο στάδιο δεν ήταν καθόλου δημοφιλή απόφαση, γι' αυτό την απέφυγε με αποτέλεσμα να μα χτυπήσει η κρίση πολύ πιο έντονα. Ε, άλλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό επηρεάζει τις καλλιέργειες. Ε, ή δημιουργούνται μερικές φορές φαινόμενα υπερπαραγωγής. Αν ε, εντοπίσουμε από την αρχή την υπερπαραγωγή, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη σταθερότητα, περιορίζοντάς την. Πάντως, ε, ένα λάθος που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή γεωργική πολιτική είναι ότι ενδώσαμε στις πιέσεις και στην, ε, στην επίδραση του Συμβουλίου και της Επιτροπής ώστε να περιορίσουμε τα μέσα ε, ε, επέμβασης, παρέμβασης των αγορών. Και αυτό το ότι περιορίσαμε αυτά τα μέτρα παρέμβασης ήταν λάθος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί δυσχέρανε στη συνέχεια τη σταθεροποίηση των αγορών. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τους καλεσμένους ε, για τη μελέτη που μας παρουσίασαν. Και χαιρόμαστε και με την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η μελέτη είναι ενδιαφέρουσα και θα ήθελε να έρθει σε επαφή με τους εμπειρογνώμονες για να ευαθύνει σε ορισμένες πτυχές και να χρησιμοποιήσει κάποιες ε, προτάσεις και για τις υφιστάμενες διατάξεις αλλά και για τη μελλοντική διαμόρφωση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Γιατί θα φτάσουμε σχετικά γρήγορα και σε αυτή την ανάγκη της αναθεώρησης. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ για την εκπόνηση της μελέτης, ευχαριστούμε για, τις ευχαριστούμε για την παρουσίαση της μελέτης και ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία μας. Proszę Państwa, mogli przechodzić do punktu 5. Αργά αλλά σταθερά λοιπόν προχωρούμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 5, την παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, της Άγκρη, την παρουσίαση λοιπόν για την κατάσταση ως προς τις πρόσφατες και επικείμενες κατεξουσιοδότηση πράξης. Wiemy, że te akty wiele οι κατεξοδότηση πράξεις ε, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά, γύρουν αμφιβολίες, μερικές φορές μας ευνηδιάζουν. Γι' αυτό και εκτιμούμε ιδιαίτερα στην ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Και μάλιστα όσο πιο νωρίς γίνεται, αυτή η ενημέρωση τόσο το καλύτερο. Σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο κύριος Γιάννης Χάπς από τη Διεύθυνση ΓΑΜΑ της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας ε, από την Διεύθυνση Κοινή Οργάνωσης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων. Μετά την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσω την ευκαιρία στους συναδέλφους για να υποβάλουν ερωτήσεις. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Σχάπ, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσουμε το πού βρισκόμαστε με τους επερχόμενους κατεξουσιοδότηση κανονισμούς. Γνωρίζετε ότι πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο που έχουμε επιτελέσει και έχουμε ενδιαφέρον να εξετάσουμε το έργο μας αυτό, την εργασία μας αυτή, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίως μας απασχολούν οι οργανώσεις, οι κοινέ οργανώσεις αγορών. Και στόχος μας είναι να μεταφέρουμε τις υφιστάμενες διατάξεις σε νέες κατεξουσιοδότηση πράξεις. Πρώτο βήμα για μας ήταν ότι καλούμεθα να ευθυγραμμίσουμε 200 κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις νέες διατάξεις της Συνθήκης Λισαβόνας και έχουμε περίπου 200 κατεξουσιοδότηση κανονισμούς και 200 αριθμιστικούς κανονισμούς. Βεβαίως δεν είναι επιθυμητά τόσο υψηλά νούμερα. Γι' αυτό εξετάσαμε τις ενδεχόμενες δυνατότητες να επανείδουμε και να συγχρονίσουμε το ρυθμιστικό αυτό έργο και να το ευθυγραμμίσουμε με τις νέες διατάξεις. Με στόχο την απλοποίηση, αύξηση της συνοχής, μείωση των ποσοστών σφαλμάτων και μείωση της γραφειοκρατικής επιβαρύνσεως. Σημαντική είναι και η πτυχή της ευθυγραμμίσεως στην ε, προσπάθεια αυτή. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν επίσης να αυξήσουμε την ασφάλεια δικαίου και να κάνουμε πιο ευανάγνωστη την νομοθεσία μας, πιο εύχριστη για τους άμεσα ενδιαφερομένους και αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι ο κυριαρχικός μας στόχος Εν τέλει, θέλουμε στο τέλος της διαδικασίας αυτής να φτάσουμε σε 20 περίπου κατεξουσιοδότηση και 20 ρυθμιστικούς κανονισμούς οι οποίοι θα καλύπτουν όλες τις κοινέ οργανώσεις αγορών στη βάση των διατάξεων που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Γεωργίας για την ενεργό συμμετοχή σας και τον πολύ ενεργό ρόλο που παίξατε. Ε, με τη συμμετοχή σας στις ομάδες εμπειρογνωμόνων κλπ. Αντιλαμβανόμεθα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε δυνατόν. Αλλά με την ευκαιρία που μου δίνετε θα ήθελα να, να ευχαριστήσω για την προσπάθεια σας αυτή. Ε, από καιρούς καιρών έχουμε συμφωνήσει ότι θα ερχόμαστε σε επαφή με τον εισηγητή και την ομάδα του, πρόκειται κ. στην περίπτωση αυτή και νομίζουμε ότι μπορούμε να ωφεληθούμε και εμείς από την εμπειρία και την εμπειρογνωσία των βουλευτών σας για να προχωρήσουμε στην διαδικασία. Υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο να συνεννοηθούμε και διμερός για την παροχή περαιτέρω εξηγήσεων. Η ομάδα μου είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για συζητήσεις και για πιο συγκεκριμένα ζητήματα που έχετε και θέλετε να συζητήσουμε. Ας έρθουμε τώρα στο πού βρισκόμαστε, ποια πρόοδο έχουμε επιτελέσει και για να ανακεφαλαιώσω έχω να σας πω ότι έχουμε ενημερώσει για τη γραμματεία σας και για τους ευρωβουλευτές σας σχετικά με τα τελευταία ζητήματα πρόοδου για το πρόγραμμα ευθυγραμμίσεως. Έχουμε και ένα σχετικό πίνακα στο τέλος του εγγράφου μας. Θα δείτε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος τους τελευταίους μήνες από τότε δηλαδή που εκδόθηκε το τελευταίο μας έγγραφο που ήταν τέλη Απριλίου. Αλλά μάλιστα και τους τελευταίους δύο μήνες μπορέσαμε να εκδώσουμε τέσσερις κατεξουσιοδότης κανονισμούς, τους οποίους έχουμε διαβιβάσει στους νομοθέτες, στους συνομοθέτες, δύο συνομοθέτες δηλαδή, για την ε, εξέταση, αφενός για τις ε, αποθηκεύσεις, αφετέρου για την έκδοση αδειών. Επίσης τρίτο, το, τα εθνικά προγράμματα στήριξης για το κρασί και τέλος sugar value sharing, κανόνες δηλαδή για τον καταμερισμό της αξίας για τη ζάχαρη στη βάση κατεξουσιοδότηση κανονισμού που έχει διαβαστεί σε εσά και εξέταση. Έχουμε και έναν αριθμό σημαντικών κατεξιοδότησης κανονισμών που βρίσκονται, ή πράξεων, που βρίσκονται στον αγωγό, όπως λέμε, δηλαδή θα έλθουν τους επόμενους μήνες και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να τους ολοκληρώσουμε και πριν από το τέλος του έτους. Ιδίως η, η κατεξουσιοδότηση πράξη για οπωροκυπευτικά επίσης για τους μηχανισμούς εμπορίου, τρίτο για την ταξινόμηση των σφαγείων, τέταρτο για ορισμένα ζητήματα μηχανισμών εμπορίου και τέλος για τα σχολικά προγράμματα, για τα προγράμματα δηλαδή για τη διάθεση γεωργικών προϊόντων στη σχολεία. Αυτά τους τελευταίους μήνες. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι είμαστε πεπισμένοι ότι Όλα αυτά θα φτάσουν στα γραφεία σας μέχρι το τέλος του 2016. Για να ολοκληρώσω την εικόνα, επιτρέψτε μου να πω ακόμη ότι μπορέσαμε να ε, χαρακτηρίσουμε ως κανονισμούς που έχουν εκπνεύσει πλέον, είναι δηλαδή πλέον εκτός ισχύω ορισμένους, και είναι σαφές ότι θα συνεχίσουμε να, εξετάσουμε, να εξετάζουμε αν υπάρχουν και πρόσθετες δυνατότητες να μειώσουμε τον αριθμό των πράξεων εφόσον αυτές οι πράξεις, οι κανονισμοί περιέχουν ρήτρες λήξεως sunset clauses δηλαδή. Αυτά σχετικά με τις διάφορες κατεξουδότητες πράξεις. Στα χέρια σας είμαστε τώρα. Εάν επιθυμείτε να θέσετε ερωτήσεις, μπορείτε να μας απευθύνετε ερωτήσεις και για συγκεκριμένα πράγματα. Για μας είναι όλα αυτά σημαντικά, αλλά για σας σίγουρα έχουν ενδιαφέρον κάποια άλλα και κάποια άλλα λιγότερο. Ευχαριστώ κύριε Σαντρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εάν με επιτρέπετε, θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της ίνοκαλλιέργειας, της αμπελοκαλλιέργειας. Ε, το καλύπτει το έγγραφό σα και αυτό και ήδη μα είπατε κάποια πράγματα. Τον Μάρτιο, όταν είχαμε συζητήσει με την Επιτροπή και είχαμε θέσει ερωτήσει, και αυτό επιτρέπει να τα δούμε με κάποια απόσταση τα θέματα και να επιστρέψουμε, νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχουμε κάποια από τα κείμενα που έχει σκοπό να τροποποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να έχουμε μια συνολική έποψη του τι επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτόν τον τομέα επί της ουσίας του θέματος, που είναι μη τι άλλο ευαίσθητος, θα πρέπει να επιμείνουμε στο ότι ό,τι και αν προταθεί να μην διαταράξει την μεταρρύθμιση του 2008, ούτε την γενικότερη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2013. Σημαντικό είναι να θυμηθούμε εδώ και να το πούμε και με σαφήνεια ότι πρέπει να διατηρηθεί το σύνολο των κανόνων που είναι εξειδικευμένοι για αυτόν τον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας και ε, τον ίνο παραγωγικό. Να παραμείνουν όλοι αυτοί οι κανόνες που ε, διασφαλίζουν τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις και την ε, σήμανση των προϊόντων στο κείμενο. Αυτά νομίζω ότι είναι ένα διάσπαστο σύνολο. Επίσης σημαντικό είναι να μην μειωθεί η, η πρόσβαση στους κανόνες για τους ενδιαφερόμενους του τομέα, για τους δραστηριοποιούμενους και σε επίπεδο γεωγραφικών ενδείξεων, οπωσδήποτε οι κανόνες πρέπει να ε, διατηρηθούν ανέπαθοι στο σημερινό πλαίσιο, ό,τι πρόταση για μας προτείνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως εισηγητής θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κόρτ, τον Γενικό Διευθυντή και τις ομάδες των συνεργατών του για τον ποιοτικότατο διάλογο που είχαμε. Να θυμίσω στις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες ότι η Γραμματεία δεν γνωρίζει πάντοτε τους κοιόδους εισηγητές που θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί μου από το συγκεκριμένο ε, κειμένου, οπότε για την ώρα αισθάνομαι κάπως μόνος. Πάντως, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποιότητα του διαλόγου που είχαμε ως τώρα. Σήμερα έχουμε τέσσερα κείμενα, τα οποία μας έχουν αποσταλεί στο Κοινοβούλιο για να εξετάσουμε, κατά εξουσιοδότηση πράξη για τις ιδιωτικές παρεμβάσεις, απλούστευση σε σχέση με τις με τους σημερινούς κανόνες και από το Συμβούλιο ε, κέντρο στην ομοφωνία, μόνο δύο χώρες ε, ξέπρασαν ενδιασμούς. Σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο, ε, τα εσωτερικά ε, σχόλια δεν ε, περίχαν καμία αντίρρηση. Έπειτα, κατά εξουσιοδότηση πράξη για τα πιστοποιητικά ε, για το όλο σύστημα της πληροφορικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναπέμπεται ε, ένα μέρος της διαχείρισης πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να παρακολουθούν το τι γίνεται στην αγορά. Να θυμίσω ότι σε προηγούμενη συζήτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον η Επιτροπή Γεωργίας, είχε εκφράσει την επιθυμία, για να μην πω την απέτηση, να διατηρηθεί η διαχείριση δεδομένων όσο έχει για να μπορούμε να προλάβουμε τις εξέλιξεις στην αγορά όταν προσπαθούμε να ορίσουμε νέους προσανατολισμούς για τις πολιτικές μας. Τρίτη πράξη, κατεπίγουσα δράση για τον τομέα των εδώ μπορεί να συνεχίσει να ισχύει ε, ο κανονισμός που ήδη υπάρχει, αλλά με μείωση των χαρτοφυλακίων και αν δούμε τις ποσότητες χώρα με περιθώριο ελιγμού 3.000 τόνους, που η κάθε χώρα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα, αυτό ευτυχώς βρήκε σύμφωνο το Συμβούλιο και μετά τελευταία πράξη για το τομέα τη ζάχαρης. Στον κλάδο αυτό θα ήθελα να σταθώ λίγο, διότι το κείμενο που μας προτείνεται αποτέλεσε αντικείμενο των διακομματεύσεων. Θέλω να τονίσω ότι το Κοινοβούλιο θα προσέξει σχολαστικά να γίνει σεβαστή πολιτική συμφωνία που είχε περάσει. Η Γενική Διεύθυνση Άγκρη, ε, μάλλον όχι η Γενική Διεύθυνση Άγκρη, αλλά αλλού, ε, σε άλλε γενικέ διευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιοι διευθυντέ προσπαθούν μέσω τη νομοθετική διαδικασία να ανακτήσουν αυτά που απόλυσαν τη στιγμή τη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν θα υπαναχωρήσει στι ε, αρμοδιότητε και τα προνομιά του και τι πολιτικέ γραμμέ που τόσο ξεκάθαρα έθεσε. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέ σε όλου και να πω ότι η Γενική Διεύθυνση Άγκρη είχε την ε, αμέριστη στήριξη του Κοινοβουλίου στη συζήτηση αυτή, ενώ εσωτερικώς υπήρχαν και άλλες διαπραγματευτικέ γραμμές. Εμείς όμως θελήσαμε να διατηρήσουμε ανέπαφο το πνεύμα της πράξης που αφορούσε τη ζάχαρη και εδώ θα μας έρθουν σύντομα δύο κείμενα. Ένα για το κρασί, ε, για τον Ινό, όπως είπαμε εδώ επανειλημμένως και στο παρελθόν, δεν μπορούμε να δεχτούμε να τεμαχιστεί, διατεμαχιστεί όλη η συζήτηση για τον Ινό, ε, για το κρασί. Δυστυχώς είναι πολλά τα διαφορετικά άτομα που ασχολούνται με τα διαφορετικά θέματα. Θέλουμε όμως ό,τι αφορά την ταυτοποίηση, είτε γενικές, είτε γεωγραφικέ ενδείξει, είτε παραδοσιακέ μέθοδοι, είτε παραδοσιακά προϊόντα, αυτά να ε, εκφραστούν ξεκάθαρα για να μην υπάρχει παραμικρή, το, παραμικρό, παραμικρή, το παραμικρό κενό στην νομοθεσία. Και για τα απορροκεπευτικά, όπως έχει προχωρήσει η συζήτηση, βλέπουμε να έχουν γίνει πολλές παρατηρήσεις από τους ίδιους τους ε, φορείς του ε, με του κλάδου και να έχουν ληφθεί και υπόψη. Ευχαριστώ για αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την θέση σε εμπορία ή το ρόλο των συντελεστικών οργανώσεων στην υλοποίηση του προγράμματος. Αυτά όλα πρέπει να αποσαφενιστούν. Διότι για να χτιστεί αυτή η ΚΟΑ Ακούγαμε καθόλου την προσπάθεια οργάνωση ότι οι συνεταιριστικέ οργανώσει είναι σημαντικέ για την προστασία των παραγωγών. Όμω από τη μεταρρύθμιση του γάλακτο και την υλοποίηση του άρθρου 122 υπάρχει μια μεταστροφή στη Γενική Διεύθυνση Άγκρη που λέει ότι πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό κείμενο για τι συνεταιριστικέ οργανώσει διότι αυτό που είχαμε για τη ΣΚΟΑ δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει εδώ να υπάρξει μια γενικότερη αποσαφήνιση. Ε, ναι. Ο κύριος Ντέση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ο κύριος Νταντάν έφτιαξε ορισμένα ε, επίκαιρα θέματα και χαίρομαι πολύ που ο συζητητής θα παρακολουθεί επί του συστήματος μια παρατήρηση. Νομίζω ότι οι κατεξουσιοδότητες συνφράξεις ορθώς ρυθμίζονται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Γίνονται δηλαδή ισχυρές έχουν επομένως ισχύ εφόσον δεν υπάρξει ένσταση από πλευράς Κοινοβουλίου ή Συμβουλίου. Άρα δεν χρειάζεται να προβληθεί ένσταση και από το Κοινοβουλίο και από το Συμβουλίο, αρκεί ένα εκ των δύο αυτών οργάνων να προβάλλει ένσταση. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο για την εφαρμογή των κατεξουσιώτησης πράξεων είχαμε υποβάλει, είχαμε μάλλον προβάλει ορισμένε στάσεις και γράψαμε έτσι κοινοβουλευτική ιστορία και μας επέτρεψε αυτό να έρθουμε και σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που τα θύμισε αυτά κ. Δαντά, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί δια της μεθόδου των κατεξουσιοδότησης πράξεων να περάσει ορισμένα πράγματα όπου πολιτικά δεν έχει καταφέρει να τα περάσει. Θέματα που ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έρχομαι και διαβάζω ξαφνικά σε έγγραφο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προωθεί διακατεξουσιοδότηση πράξεως. Για παράδειγμα, στον παράγοντα 0,3 για την καλλιέργηση ε, ε, ε εδαφών είδαμε ότι δεν έγινε σεβαστό αυτό και προτάθηκε το 0,7 της 0,7 ως παράγον, ως συντελεστής δηλαδή. Οφείλουμε βέβαια να ζήσουμε με τις κατεξουσιαδότητες συμπράξεις και εάν είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαπιστώνω ότι είναι διατεθειμένη, μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτήν και για τα θέματα των κατεξουσιοδότησης πράξεων και υποφελία βεβαίω των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Αγγιλέρα, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα ευκαιρία της συζήτησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφερθώ σε κάτι που άπτε περισσότερο των αρμοδιοτήτων της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, όχι τόσο της Άγκρη, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να το επισημάνουμε στην Επιτροπή μας. Τον περασμένο Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία πρόταση για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγιας 2029 ε, για την ασφάλεια των φυτών. Και μάλιστα φαίνεται ότι θα υποβληθεί για ψηφοφορία τέλη Ιουνίου. Αυτή η τροποποίηση της οδηγίας, η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας, αποδυναμώνει τους φυτογενομικούς ελέγχους για να αποφύγει την εισαγωγή ε, ασθενειών ε, σημαντικών που θα βλάψουν τα εσπεριδοειδή. Προτείνεται χαλάρωση των ελέγχων για ε, αρρώστιες όπως το black spot και ένας καρκίνος των εσπεριδοειδών. Νομίζω ότι θα πλήξουμε τον κλάδο προκυπευτικών με την εισαγωγή μολυσμένων εσπεριδοειδών που μπορεί καλύτερα να φτάσει στις ε, ευρωπαϊκές ζώνες παραγωγής. Από τη στιγμή που έχουμε εσωτερική αγορά, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν πια έλεγχοι, ώστε από τη στιγμή που θα εισαχθεί το μολυσμένο φυτό θα κυκλοφορήσει. Είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαλαρώνει του κινδύνου για αρρώστιε ε, των φυτών, εμπροκειμένου των εσπεριδοειδών και μάλιστα τροποποιώντα ένα παράρτημα τη οδηγία 2000 κάθετο 29. Ήδη ε, είδα ότι η ημερομηνία της απόφασης αναφέρει την 11η Μαΐου ε, και τη δημοσίευση στις 13 Μαΐου στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί προβλέπονται ε, τα σχετικά κριτήρια και μάλιστα προσωρινά, όχι μόνιμα, μέχρι το 2019 αρχικά. Με την τροποποίηση, με την πρόταση τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μονιμοποιεί αυτό το πρώην προσωρινό μέτρο. Αυτό είναι απαράδεκτο να χαλαρώνουμε τους ελέγχους στις εισαγωγές προϊόντων και μάλιστα για τόσο σημαντικές αρρώστιες των φυτών όπως είναι ο, ο καρκίνος των εσπεριδοειδών ή το black spot στα εσπεριδοειδή. Και μάλιστα από τη στιγμή που ξεκινήσαμε από εδώ θα μπορούσαμε να επεκταθούμε και σε άλλα θέματα. Είναι αδιανόητο με τη δικαιολόγηση ότι κατευθύνονται στη βιομηχανία αυτά τα προϊόντα, χαλαρώνουμε τους κινδύνους και έχουμε και μία άλλη αρρώστια το, μαστοσ... το μαστοστίβια λεοκοτρέτα. Αναφέρεται πραγματική θεραπεία μόνο όταν σε όλες τις χώρες προβλέπεται ψυχρό θεραπεία των προϊόντων. Δεν ξέρω ποιο στόχο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαλαρώνοντας τους κινδύνους ε, ε, στις εισαγωγές ε, σπεριδοειδών. Απ' τη μια χαλαρώνουμε τους κινδύνους και αφήνουμε ξέφραγο αμπέλη για τις ασθένειες των φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά διαρριγνύουμε τα αιμάτια μας όταν μας χτυπάει μια τέτοια αρρώστια. Ποια είναι η επιχειρηματολογία της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ ε, για την χαλάρωση αυτού του κίνδυνου. Είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διάβημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εδώ σοβαρό πρόβλημα με τη μαύρη κοιλίδα και τον ε, καρκίνο των εσπεριδοειδών. Πώς είναι δυνατόν ενώ είχαμε αποφασίσει προσωρινά μέτρα να τα μονιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την τροποποίηση των παραρτημάτων. Είναι απαράδεκτο να χαλαρώνουμε έτσι τους ελέγχους των εισαγωγών και δεν ξέρω ποιον εξυπηρετούμε με τέτοια αποδυνάμωση των ελέγχων. Ευχαριστούμε κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, και εγώ ήθελα να λάβω το λόγο για αυτό το θέμα των τη πράξεων, αλλά οι συνάδελφοι είπαν ήδη κάποια στοιχεία που θέλω και εγώ να αναπτύξω, κυρίως ο κ. Νταντά και Αντριέ. Ήθελα να υπογραμμίσω ότι Κάποιε φορέ δεν γνωρίζουμε όλε τι πτυχέ επακριβώ από την αρχή και μετά έχουμε πολύ χρόνο για να αντιδρώσουμε. Αλλά τώρα θα ήθελα να σταθώ στην κατεξόδηση πράξη για τα προκυπευτικά, διότι έχουν γίνει κάποια βήματα πρόοδου, είναι σαφέ και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τη Γενική Διεύθυνση Άκρη. Αλλά εύχομαι η τελική πράξη που θα, που θα επιβεβαιώσει αυτά τα θετικά βήματα θα είναι πραγματικά πιστή στην εκδοχή που τώρα έχουμε δει. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλους ε, ομιλητές στον κατάλογο. Οπότε στρέφαμε προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Σχάπ, και το ρωτώ αν θέλει να ξαναλάβει το λόγο για να απαντήσει. Θα του είμαστε ευγνώμονες αν το έκανε. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. όλοι έχουμε ακριβώς την ίδια μέρημνα. Να προχωρήσουμε στο το δυνατόν πιο ομαλά με όλο αυτό το εγχείρημα. Και θα επαναλάβω κάτι που έχουμε πει επανειλημμένω. Νομίζω η αίσθηση αυτή επικρατεί και εδώ, στο Κοινοβούλιο. Ότι ως τώρα η συνεργασία μας έχει πάει καλά. Βεβαίως, πέραν αυτού, περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν πάντοτε. Γνωρίζω ότι η μια ή η άλλη πρωτοβουλία μπορεί να φαίνονται πιο περίπλοκες από άλλες, όπως για τα απορροκυπευτικά. Αυτή η πράξη φαίνεται να σας αποσχολεί πολύ, πολλούς από εσάς. Οπότε σας προσκαλώ μαζί μας να καθίσουμε όλοι μαζί και να κοιτάξουμε την ουσία του ζητήματος, την αυτό που πιο πολύ σας προβληματίζει. Επίσης, πιο συγκεκριμένα, είναι επίσης αθές, όπως είπε ο κύριος Αντριέ, και εξ όσων κατάλαβα, το θέμα είναι οι κανόνες εμπορίας για τον ίνο. και τις διαδικασίες επισήμανσης. Εδώ έχουμε μια λίγο διαφορετική προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι η σχετική πρόταση θα είναι πολύ γρήγορα, αλλά εάν δούμε το χρονοδιάγραμμα, αυτό είναι στο τμήμα 5, λοιπές πρωτοβουλίες, όπου θα γίνει στο προσεχές μέλλον αυτό, αλλά προτού προτείνουμε το οτιδήποτε θα υπάρξει μια διαδικασία αξιολόγησης Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες και συγκεκριμένα υπάρχουν αντιδράσεις από τον ίνοπαραγωγικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε προσεκτικότατα. Για τα υπόλοιπα στοιχεία πρέπει να έχουμε μία κοινή κατανόηση, μια συμφωνία και πολιτική και όπως είπαν κάποιοι βουλευτές ο σκοπός δεν είναι να επανερμηνεύσουμε τις βασικές πράξεις. Δεν είναι καθόλου αυτή η πρόθεσή μας. Θέλουμε απλώς να εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία και όπως υπόθηκε, ο νόμος έχει αποτυπωθεί στους βασικούς κανονισμούς. Οπότε, η λογική μας είναι ότι δεν αγγίζουμε τους βασικού κανόνες, αλλά με κατεξουσιοδότηση πράξη φροντίζουμε να προσαρμόσουμε τους κανόνες στο πνεύμα που θέλαμε να έχουν αυτοί. Και αυτό έχει οδηγήσει ως τώρα τη δουλειά μας. Είμαι βέβαιος ότι επιτυχώς θα συνεχίσουμε σε αυτή την άγουσα. Η κυρία Καρσία έθεσε μια ερώτηση ιδίως για την όσο black spot και είπατε νομίζω ορθώς κι εσείς ε, ότι πρέπει να ληφθεί με έρημνα, όμως δεν είναι δυστυχώς η δική μου ειδικότης, Εάν με επιτρέπετε να μεταφέρω τα σχόλια σας στη Γενική Διεύθυνση Σάντε και ελπίζω ότι την επόμενη φορά που θα είναι εδώ θα μπορέσουν να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ως προς την κάλυψη των συγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων, εγώ είχα ε, πάει σε επίσκεψη σε συγκεκριμένες περιοχές. Βλέπω γύρω μου ότι δεν έχω συναδέλφους να μου κάνουν εννοήματα ότι κάτι ξέχασα από όσα είδαμε που είναι πολύ σημαντικό. Ε, και από όσα ρωτήσατε, πάντως σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και είμαι στη διάθεσή σας για να επιστρέψω όποτε με χρειάζεστε. Σας ευχαριστούμε. Σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. γιατί ε, χαίρομαι που πεθυμίσατε ότι κρατούμε το, τηρούμε το πνεύμα του κανονισμού ε, των γενικών διατάξεων για τις της πράξης. Αυτό το πνεύμα όμως με ανησυχεί κάπως, γιατί μερικές φορές ε, μας ξεφεύγει το πνεύμα. Είναι κάπως άειλο. Εν πάση περιπτώσει, αστείευομαι. Σίγουρα θα συνεχιστεί η συζήτηση και η συνεργασία μας και επ' ευκαιρία της συζήτησης έκθεσης ο κύριος Νταντά θα συναντηθεί με τους κοιόδη ηγητές, οπότε θα συγκεκριμενοποιηθούν πολλά ζητήματα εκεί. Πάντως, ελπίζουμε ότι θα διεκπαιρεώσουμε το θέμα αισίως. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουμε και εμεί προσδοκίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν και οι Γεωργία προσδοκίε από εμά. Και είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη τι επιθυμίες και τι προσδοκίε για τον Γιώργο. Αυτά. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη το σημείο 5. Και ολοκληρώσαμε και την απογευματινή μα συνεδρίαση, γιατί δεν έχουμε άλλα σημεία. Αύριο θα ξεκινήσουμε το πρωί στι 9 με καλεσμένο τον Επίτροπο Μιγέλα Αρίας Κανιέτε. Θα συζητήσουμε μαζί του για το ρόλο της γεωργίας στις κλιματικές αλλαγές και στο πλαίσιο όλων αυτών των προκλήσεων που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές. Αυτά, ραντεβού αύριο στις 9 παρακαλώ. Καλό σας απόγευμα.